No. Ok, mes chers collègues, Monsieur le Commissaire, je vous propose d'ouvrir notre séance. Je remercie les. Ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ τους δημοσιογράφους που παίρνουν φωτογραφίες στη συνεδρίασή μας και παίρνουν διάφορες εικόνες. Λίγη ησυχία, αν έχετε την καλοσύνη. Να επενθυμίσω ότι πρόκειται περί κοινή συνεδριάσεω τη Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων και τη Ειδική Επιτροπή ε, για ε, Φορολογικά Έσοδα. Οι δύο επιτροπέ θέλαν να διεξαχθεί από κοινού η ακρόαση του Επιτρόπου του κ. Μοσκοβίση. Ευχαριστώ τον Επίτροπο που δέχτηκε να έρθει για να μας ε, παρουσιάσει το κείμενο που υφετήθηκε κατόπιν προτάσεώς σας στις 18 του περασμένου Μαρτίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, να, και ότι απάντησε και στις ερωτήσεις των ε, εισηγητών μας και των μελών. Θα είδατε την ημερήσια διάταξη της κοινής αυτής συνεδριάσεως που περιορίζεται στην ακρόαση του Επιτρόπου. Αν δεν έχετε σχόλια, θεωρούμε συγκεκριμένη την ημερήσια διάταξη να υπενθυμίσω ότι ο σύμφωνος κανόνας της Επιτροπής μας αυτή η συνεδρίαση είναι δημόσια και μεταδίδεται και μέσω διαδικτύου. Δίνω το λόγο στον Πρόεδρο τον κύριο Φέρμπερ όσον αφορά την Οικονομική και Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ, αλλά θα ήθελα να καλωσορίσω, να πω μάλιστα ε, συγγνώμη εξ ονόματος του Προέδρου μας, του κυρίου Γκουαλτιέρη, ο οποίος θα έρθει κατά τη διάρκεια του απογεύματος, για τη δική μας Επιτροπή Οικονομική και Νομισματική έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτή η κοινή ακρόαση με τον Επίτροπο Μοσκοβισή. Σας καλωσορίζω λοιπόν και εγώ θερμότατα εξ ονόματος Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Θα ήθελα μόνο να πω το εξή. Πρώτον, γιατί περί αυτού πρόκειται σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε μία πρόταση για ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις φορολογικές συμφωνίες. Η δική μας Επιτροπή ΕΚΟΝ έχει την αρμοδιότητα για τα φορολογικά ζητήματα. Οπότε αυτή τη στιγμή οριστούν οι εισηγητές θα ασχοληθούμε και με την νομοθετική πτυχή της πρότασης αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τότε θα αρχίσει αυτή η δουλειά, εξού και είναι κοινή ακρόαση. Δεύτερον, στην Επιτροπή μας, ΕΚΟΝ, αναθέσαμε μία νομοθετική έκθεση πρωτοβουλίας, Νίτερ Μάγερε είναι οι συγητές μας και σε αυτή την έκθεση θα βασιστούμε και στα πορίσματα της Επιτροπής Τάξη αυτής της Ειδικής Επιτροπής ε, και θα προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει προτάσεις για νέα νομοθετική πρωτοβουλία. Γι' αυτό, για να εξηγήσω για ποιο λόγο γίνεται από κοινού η ακρόαση, σας ευχαριστώ πολύ για τη διεξαγωγή αυτή και αγαπητέ Αλάν, θέλω να σε ευχαριστήσω και σένα για την αγαστή συνεργασία που έχουμε οι δύο επιτροπές. Σου ξαναδίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και Μάρκο, Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Αντιπρόεδροι, κυρίες και κύριοι αξιότιμο μέλη της Επιτροπής, έχω την εντύπωση ότι είμαι ο πρώτος ε, που έρχομαι εδώ στην ειδική μεικτή επιτροπή για μια ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με την φορολόγηση των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Έγινε μια συζήτηση την περασμένη εβδομάδα όπου τοποθετήθηκα και είπα πως Κατά τη γνώμη μου είναι λίγο ανησυχητική η κατάσταση σε σχέση με τη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Σε μεγάλο βαθμό είναι ανοιχτή η οικονομία και η έλλειψη συντονισμού των πολιτικών και των φορολογικών κανόνων των κρατών μελών δημιουργεί πλέον ε, θεμελιώδη προβλήματα για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι δεν είναι, υπάρχει ομοιομορφία, διαφάνεια και άρα ούτε και αποτελεσματικότητα σε αυτό το σύστημα. Ας μην ξεχνάμε ε, ότι οι επιχειρήσεις δημιουργούν το πλούτο και έτσι οι διαφορετικοί φορολογικοί κανόνες οδηγούν σε κατάτμιση της ενιαίας αγοράς ε, και είναι εξαιρετικά ακριβό πλέον για τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με τις πολύ διαφορετικές νομοθεσίες που υπάρχουν. Αντιμετωπίζουν λοιπόν φραγμούς που αναχαιτίζουν και την ανάπτυξή τους, ε, εμποδίζοντάς τους να μας βοηθήσουν ώστε να αντεπεξέλθουμε και στις μεγάλες προκλήσεις σημερινής αποχής. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις κυβερνήσεις είναι η συλλογή των φόρων, ε, το πρόβλημα, το βασικότερο πρόβλημα είναι η, επιθετική, ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός ε, που οδηγεί στην αξιοποίηση αυτών των ε, ανακολουθιών και των διαφορών που υπάρχουν ανάμεσα στα εθνικά φορολογικά συστήματα. αυτό το εκμεταλλεύεται τα επιχειρήσεις, ταυτόχρονα είναι μια κατάσταση ανυπόφορη για τους πολίτες που καλούνται να δώσουν εκείνη την απάντηση στην οικονομική κρίση. Σε σχέση τώρα με την κυριαρχία και τον φορολογικό ανταγωνισμό καταλήγουμε σε μια φορολογική μειοδοσία ε, και δεν λαμβάνονται υπόψη άλλοι κανόνες, ε, ε, ιδίως στη δημοσιονομική, παραδείγματος χάρη, επιδίδονται οι επιχειρήσεις, οι μεγάλες επιχειρήσεις ε, σε φορολογικό και τα κράτη σε φορολογικό ανταγωνισμό και τελικά αποφασίζουν οι επιχειρήσεις ε, πώς θα φορολογηθούν και όχι πλέον τα κράτη. Είναι άδικο αυτό το σύστημα και είναι υποφελές ε, για τους ισχυρότερους εις βάρος όλων των υπολείπων. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι διαβρώνεται το ίδιο το ε, η ίδια η κοινωνική συμφωνία ανάμεσα στους πολίτες ε, και του, τα κράτη. Δηλαδή η χρήση της φορολογίας για την χρηματοδότηση των κρατικών ε, λειτουργιών. Θα πρέπει λοιπόν τα, ταχύτατα να αναλάβουμε μία δράση μεγάλης εμβέλειας και μπορώ να σας πω ότι παρότι είναι ρηξικέλευτο το πακέτο διαφανές που εγκρίθηκε πριν από δύο εβδομάδες δεν θα πρέπει να σταματήσουμε εκεί. Ε, συμμορφούμενοι ούτω ή άλλω και με τους στόχους του Κοινοβουλίου. Δηλαδή να ανακτήσουμε την αξιοπιστία μας ε, ε, αντιμετωπίζοντα το φορολογικό ανταγωνισμό των κρατών μελών. Έχουμε μια μελλοντοστραφή πολιτική, μια ενιαία πολιτική, ένα προβλέψιμο διαφανέ πλαίσιο για τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να ανακτήσει και η αξιοπιστία στα μάτια των πολιτών μας. Η φορολογία θα αναδειχθεί σε προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα το ξεκαθαρίζω ότι η ανάπτυξη και η απασχόληση είναι οι βασικότερες ύψιστες προτεραιότητες του τωρινού νομοθετικού πακέτου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το σχέδιο δράσης ε, της Επιτροπής για να υλοποιηθεί προϋποθέτει ότι θα αναλάβουν δέσμευση τα κράτη-μέλη διότι ε, όπως ξέρετε εκείνοι αποφασίζουν, τα κράτη-μέλη αποφασίζουν ε, και για να εκδοθεί μια οδηγία απαιτείται ομοφωνία. οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι αυτό αποτελεί τροχοπέδι χρειάζεται ε, μία ευφυής ισορροπία ε, δυνάμεων ανάμεσα στα θεσμικά όργανα αλλά και την πίεση των πολιτών ώστε να κινητοποιηθούν τα κράτη-μέλη. Είμαι πεπισμένος ότι θα είναι φιλόδοξες οι λύσεις οι οποίε θα καταλήξουν τα κράτη-μέλη λύσεις που ήδη προτείνουμε εμείς από πλευρά της Επιτροπής και που θα προτείνουμε και στο μέλλον. Σας είπα ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε στο πακέτο της διαφάνειας και σας είπα ότι είναι επαναστατικό το πακέτο. Να σας εξήγησω γιατί. Ε, η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τα tax rulings, παραδείγματο χάρη, είναι σημαντικότατο πρώτο βήμα, ούτω ώστε να είναι διαφανέστερο και δικαιότερο το φορολογικό περιβάλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα παραμένει ένα βήμα, το πρώτο βήμα. Θα ακολουθήσουν και άλλα από πλευρά τη Επιτροπή και των κρατών μελών. Είναι απαραίτητο λοιπόν να ενισχύσουμε το νομοθετικό πλαίσιο τη φορολογία στην Ευρώπη και να ε, μετέλθουμε των απαιτουμένων μέσων, ώστε να έχουμε ένα αποτελεσματικό τροφολογικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α περάσω σε πιο πρακτικέ πληροφορίε σε σχέση με το πακέτο διαφάνεια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βασικότατο στοιχείο αυτού του πακέτου είναι η πρόταση που κάναμε σε σχέση με την ανταλλαγή πληροφοριών για τα tax rulings. Ξέρετε τι πρόκειται θα είναι στη διάθεση όλων των κρατών μελών πληροφορίες ε, σε σχέση με τις επιπτώσεις που έχουν αποφάσει των άλλων κρατών μελών στη δική τους ε, φορολογική βάση. Είναι απλή η λειτουργία, βασίζεται στην ε, διοικητική συνεργασία για τους άμεσους φόρους. Έτσι, υπάρχουν, έτσι έχουμε ένα πλάσιο, πλαίσιο για να συνεργαστούμε τα κράτη-μέλη σε σχέση με την φορολόγηση των επιχειρήσεων. Οι κάποιες πληροφορίες ανταλλάσσονται αυτόματα, κάποιες κατόπιν αιτήματος, κάποιες αυθόρμητα. Και βλέπουμε, επειδή έχω προσωπική εμπειρία στον τομέα, όταν ε, ζητούμε πληροφορίες, ε, παίρνουμε ή όχι μία απάντηση, μία πλήρη ή ε, μερική απάντηση ή καταλαβαίνετε λοιπόν πως ένα τυποποιημένο σύστημα ανταλλαγής ε, πληροφοριών εξασφαλίζει ε, μια πολύ καλύτερη ποιότητα. Η οδηγία προβλέπει και άλλους ε, τρόπους συνεργασίας, κοινούς, κοινές ελεγκτικές αποστολές από πλευράς των φορολογικών διοικήσεων κρατών μελών. Ε, στη συνέχεια, μετά το Δεκέμβριο του 2014 και χθε εφαρμογή τη οδηγία, ε, τι συμβαίνει. Έχουν λάβει τη δέσμευση στα κράτη-μέλη, ε, ούτω ώστε να ανταλλάσσουν αυτόματα όλε τι φορολογικέ πληροφορίε σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα του ΩΣΑ. Βλέπουμε ότι μεγάλε επιχειρήσει στην ενιαία αγορά έχουν καταλητικό ρόλο και έτσι με τον οδηγία για την διοικητική συνεργασία ε, ε, διευκολύνεται η εργασία των φορολογικών διοικήσεων. Πόρο απέχουμε όμως από μια ενοποιημένη, ένα ενοποιημένο μειόμορφο σύστημα. Πρέπει λοιπόν ε, να υπερβούμε ε, αυτό το ζήτημα των tax rulings ε, για να διατηρήσει το ρόλο του προτεργάτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον θα μπορούσε μια δυνατότητα να είναι, όπως τονίζει και το Κοινοβούλιο στην έκθεσή του για τη φορολογία, να διευρύνουμε τις υποχρεώσεις που έχουν κάποιες βιομηχανίες σε σχέση με την κοινοποίηση κάποιων οικονομικών πληροφοριών. για ε, τα κέρδη και τα μερίσματα ανά χώρα. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη στον τομέα αυτό και ε, φυσικά αντιλαμβάνεστε τον αντίκτυπο τέτοιων αποφάσεων στην οικονομική ζωή των κρατών μελών, διότι περί αυτού πρόκειται. Μία άλλη ιδέα είναι ε, η ετήσια έκθεση του ΩΣΑ ανά χώρα ε, που αναμένεται για το φθινόπωρο το 2015, βάσει τη οποία οι πολυεθνικές επιχειρήσει κοινοποιούν κάποιε πληροφορίε στι φορολογικέ αρχέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμη δεν έχει λάβει την ε, απόφαση σε σχέση με το ε, βέλτιστο τρόπο λειτουργίας ε, διότι ε, χρήζει διεξοδικότερης ανάλυση στο ζήτημα όπως σας είπα. Για να κάνουμε αυτή την ανάλυση που είναι βασική προϋπόθεση ώστε να καταθέσουμε μελλοντικά προτάσεις και να πω παρενθετικά ότι παρακολουθώ εκ του συνεγγύς και αναλαμβάνω προσωπική δέσμευση για αυτό το ζήτημα πέραν από το ρόλο μου του Επιτρόπου διότι ο στόχος μου είναι να ε, προχωρήσουμε το περισσότερο δυνατό, όχι να κάνουμε τις μελέτες για να πούμε στο τέλος «Α, κατόπιν μελέτες δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα», όχι, χρειαζόμαστε ένα κρατεό ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ε, στα, στις αρχές ε, του δεκαετία του 90 καταλήξαμε σε παραδείγματο χάρη σε ένα κώδικα διοντολογίας των επιχειρήσεων σε διακυβερνητική και θελούσια βάση λειτουργεί αυτός ο κώδικας διοντολογίας. Παρ' όλα αυτά όμως αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα διάφορων προβληματικών καθεστώτων ε, τα κριτήρια στα οποία βασίζεται ο κώδικας όμως είναι απαρχαιωμένα ε, λόγω των εξελίξεων στον φορολογικό τομέα και άρα δεν είναι αποτελεσματική η δράση μας. Ε, εξετάζουμε λοιπόν το ενδεχόμενο να αναβαθμίσουμε αυτόν τον τονίζω διακυβερνητικό ε, κώδικα διοντολογίας. Επίσης είναι σημαντικό για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα να ποσοτικοποιούμε και άρα να προσμετρούμε και τη δράση μας. Ε, συλλογή λοιπόν αξιόπιστων στοιχείων από πλευρά των κρατών μελών σε σχέση με την φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. Η Μάρκρατ Στάγκερ ε, που θα ακούσετε στην ε, η Μάργαρετ Βέσταγκη συγγνώμη την οποία θα ακούσετε ούτω ή άλλω, θα σα δώσει περισσότερε πληροφορίε ε, για, αυτό το, για αυτό το θέμα. Ε, δεν ε, θα ασχοληθώ εγώ ε, με αυτό, διότι είναι, δεν είναι άμεση αρμοδιότητα ε, για μένα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμω θα πρέπει να συνεργαστεί και σε διεθνέ επίπεδο. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με το G20 για το BEPS, δηλαδή για την αντιμετώπιση τη διάβρωση φορολογική βάσεις ε, για να υπάρχει διαφάνεια στα τρας παραδείγματος χάρη. Εδώ και χρόνια αγωνίζομαι σε αυτό το τομέα και με τα νέα ε, καθήκοντά μου θα μετάσχω άμεσα στις εργασίες του G20 σε λίγες εβδομάδες ε, διότι μην ξεχνάτε ότι έχουμε και την ετήσια συνέλευση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Θα υπάρξουν εξελίξεις λοιπόν σε παγκόσμιο επίπεδο για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών Είδατε την περασμένη εβδομάδα ότι υπογράψαμε, κυρώσαμε μια συμφωνία με την Ελβετία. Ακολουθούν Λίχτενστάιν, Άγιος ε, Μαρίνος ε, Ανδόρε ε, και ο στόχος είναι να εφαρμοστεί το διεθνής κανόνας του ΟΣΑ και του G20. Συγγνώμη αν μακρηγορά, αλλά ήθελα να έχουμε ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη συζήτησή μας. Τα κράτη-μέλη επίσης προσπαθούν να προσεγγίσουν ένα νέο πλαίσιο για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων όπου θα φορολογείται η αξία, η προσθέμενη αξία εκεί που δημιουργείται. Δηλαδή ο τόπος φορολόγησης και ο τόπος δημιουργίας του πλούτου θα τείνουν να συγκλίνουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, διότι ε, υπάρχουν περιπτώσεις ε, όπου δεν υπάρχει φορολόγηση ούτε εκεί που διαπιστώνεται δημιουργία ε, της αξίας ούτε εκεί που έχει την έδρα της η επιχείρηση. Να σας θυμίσω επίσης πέρα από αυτά τα μέτρα που προανέφερα για την ανταλλαγή των πληροφοριών υπάρχει και η οδηγία για τη μητρική θηγατρική ε, υπήρξε και μία ρήτρα για την κατάχρηση των ε, φορολογικών, ε, της φορολογικής ευελτιστοποίησης σε βάση υβριδικών φορολογικών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε γενή χαρακτηριστικά όπως το ευρώ, η ενιαία αγορά που όμως λειτουργεί βάσει 28 διαφορετικών φορολογικών συστημάτων. Κάθε κράτος έχει τους δικούς κανόνες τις δικές του προτεραιότητες και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να βασιστεί μόνο ε, στον ΩΣΑ, Θα πρέπει από μόνη της ε, να εργαστεί προς ένα ενοποιημένο ε, σύστημα. Ο Ιούνιος του 2015 είναι ο στόχος μας για την εναρμόνιση της φορολογικής βάσης, το σύστημα άξης, ούτω ώστε να έχουμε ε, μειωμένες δυνατότητες ε, κατάχρησης ε, των φορολογικών κανόνων. Αυτό για την ανταγωνιστικότητα, για τη διαφάνεια αλλά και για την ηθική έχει ιδιαίτερη σημασία. Ελπίζω λοιπόν να υπερβούμε τα, αυτά που έχουμε ήδη ανακοινώσει σε σχέση με τη διαφάνεια. Είναι απαιτή απαιτείται να, να το κάνουμε αυτό και εξάλλου περιμένουμε ότι θα εγκριθεί το σχέδιο δράσης πριν το καλοκαίρι από, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζουμε τα κράτη-μέλη να συμβάλλουν ενεργά στην προετοιμασία, στην έγκριση και την εφαρμογή του σχεδίου δράσης. Το ίδιο επιθυμώ και για το Κοινοβούλιο και είμαι ε, στη διάθεσή σας ε, να ακούσω τις ερωτήσεις σας ε, στο μέτρο φυσικά που μπορώ να σας απαντήσω. Σας ευχαριστούμε. Ήσασταν εξαιρετικά συνθετικός και σαφέστατος. Ας ακούσουμε πρώτα τους ε, ε, συνεισηγητές μας ε, για την Επιτροπή Τάξη και ΕΚΟΝ και στη συνέχεια θα ακούσουμε τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Η Ελίζα Φερέρα, συνεισηγήτρια για τις δύο επιτροπές. Ευχαριστώ, θα μιλήσω τη Δημητρική μου. Ευχαριστούμε που ήρθατε, Επίτροπε. Σας ευχαριστούμε που επιτέλους ε, εξ ονόμας Ευρωπαϊκής Επιτροπής ασχολείστε προσωπικά με αυτό το ζήτημα της καταπολέμησης φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής με την απαιτούμενη αποφασιστικότητα. Διότι είναι θέμα πλέον αξιοπιστίας ε, του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τους πολίτες όταν ζητείται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από τους πολίτες θυσίες τεράστιες διότι υπάρχει το δημοσιονομικό έλλειμμα. Ταυτόχρονα, ε, στον ίδιο ευρωπαϊκό χώρο ανεχόμαστε αυτό που συμβαίνει με τις μεγάλες επιχειρήσεις που σχεδόν δεν πληρώνουν φόρους και εκμεταλλεύονται αυτή την, αυτό το φορολογικό ανταγωνισμό. Ε, είναι πλέον απαράδεκτη, ανυπόφερη η κατάσταση. Περιμένουμε τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, με ορίζοντα τον Ιούνιο και χαιρετίζουμε τις αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί. Θα ήθελα, Επίτροπε, ε, περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά που μας είπατε σε σχέση με τις εργασίες του ΟΣΑ. Βλέπουμε ότι ε, υπάρχουν πολλά σημαντικά βήματα που απαιτούνται για να επιτύχουμε διαφάνεια και αναγνώριση των πρακτικών των πολυεθνικών επιχειρήσεων ε, κάποια από τα στοιχεία του action plan, του σχεδίου δράσης, κοινοποιούνται. Με ποιο τρόπο λοιπόν, ερωτώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προωθήσει αυτό το έργο και πώς προετοιμάζεται εφόσον ε, ε, επιθυμεί να έχει ολοκληρωμένη δράση, πώς προετοιμάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για να αντιδράσει σε σχέση με τις προτάσεις του ΟΣΑ. Και επίσης, σε ποιο βαθμό συνειδητοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι σε επίπεδο Συμβουλίου αρχίζουν ε, να κινητοποιούνται τα κράτη-μέλη που είναι στην πηγή αυτού του φορολογικού πολέμου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης θα ήθελα να ρωτήσω τι σκοπεύει να κάνει σε σχέση με τις πληροφορίες ε, του scoreboard για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Από τότε που άρχισε να επιθεί προσοχή όλων το κοινοβούλιο σε αυτό βλέπουμε μετακινήσεις των ε, ε, κεφαλαίων ως προς τις ε, ξένες επενδύσεις και βλέπουμε ότι το 2013 κατά μέσο όρο έχουν χάσει την ελκυστικότητά τους κάποια κράτη-μέλη κατά 35% παραδείγματος χαρή. Βλέπουμε ε, το Λουξεμβούργο σε αυτό το scoreboard αντίθετα να έχει ελκυστικότητα 216%. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι ασχολείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το έλλειμμα, ε, αλλά δεν λαμβάνει υπόψη αυτές τις πληροφορίες του πίνακα βαθμολογίας του scoreboard για να αποτιμήσει την κατάσταση. Εννοώ ότι υπάρχουν διεθνώς αμυντικοί μηχανισμοί από πλευράς κράτων μελών. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, θα ανταγωνιστούμε όλοι προς τα κάτω, να πληρώνουμε λιγότερο το ίδιο και επιχειρήσει, έτσι δεν θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το ελάχιστο, ε, δηλαδή ε, τι ελάχιστε υπηρεσίε που προσφέρει ένα ευρωπαϊκό κράτο ε, στου πολίτε του. Λοιπόν, υπάρχει πολιτικό πρόβλημα σε σχέση με αυτέ τι πληροφορίε. Τι μπορεί να περιμένει το Κοινοβούλιο από εσά, στο πρόγραμμα εργασία σα. Θα θέλαμε όσο το δυνατόν νωρίτερα να έχουμε στη διάθεσή μα αυτέ τι πληροφορίε. Σε ευχαριστώ Ελίζα. Όσον αφορά την ερώτηση που θέσατε για τον Όσα, θα πρέπει ο Επίτροπος να γνωρίζει ότι αύριο το πρωί θα έχουμε ακρόαση του κυρίου Γκουρία που θα έρθει με τους συνεργάτες του και κυρίως ε, όλους εκείνους που ασχολούνται με το θέμα όσον αφορά τη σημαντικό αυτό οργανισμό. Ο συνεισηγητής είναι ο κύριος Μάικλ Τόιρερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριοι Πρόεδροι και κύριε Επίτροπε. Τρεις ερωτήσεις έχω εγώ. Σας ευχαριστώ καταρχάς ε, που ήρθατε εδώ στην Επιτροπή, στην Κοινή Ακρόαση, Τάξη και Έκον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα κατέθεσε μία πρόταση πάρα πολύ φιλόδοξη για μια νέα οδηγία. Θα μπορούσατε από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αξιολογήσετε για ποιο λόγο στο μέλλον η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών θα αποτρέψει τα στρεβλά, ε, το φορολογικό ανταγωνισμό ή την επιθετική πολιτική. Και υπάρχει καμιά αντίδραση για την προηγούμενη εθελούσια ανταλλαγή και αυθόρμητη. Έχετε καμιά εκτίμηση γιατί δεν λειτουργήσε, αν δεν λειτουργήσε επαρκώς. Από τα όσα γνωρίζετε από τη σημερινή σας δραστηριότητα ως επίτροπος ή την προηγούμενη. Πού οφείλεται αυτή η κατάσταση. Έχει να κάνει με τον κώδικα συμπεριφοράς. Μήπω δεν λειτουργήσε από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ σωστά στο παρελθόν, διότι η νομοθεσία υπήρχε και προηγουμένως. Αλλά από ό,τι φαίνεται το έτο 2012 ε, υπήρξε μια ομάδα ε, για τον κώδικα δεοντολογίας όπου διαπιστώθηκε ότι δεν διαβιβάζονται στοιχεία. Πρόκειται για το Βέλγιο νομίζω τότε. Αλλά εκτό του Βελγίου νομίζω υπήρχαν και άλλες ε, συνεδριάσεις τέτοιε ή άλλε χώρε. Αυτή ήταν η δεύτερη ερώτηση. Και η τρίτη, θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια σύσταση τι να κάνουμε στο μέλλον έτσι ώστε οι Υπουργοί Οικονομικών που έρχονται στην Επιτροπή μας, άκουσα από συναδέλφους, ότι όταν προσπάθησαν στο παρελθόν να ρωτήσουν ε, ε, και να προσκαλέσουν υπουργού Οικονομικών να βάγισαν ε, και εσάς μεταξύ αυτών. Εμείς γιατί δεν τα καταφέρνουμε και έρχονται στην Επιτροπή Τάξη και όχι στην ΕΚΟΝ, μπορείτε να μας πείτε. Και για το ΦΑΤΚΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, ξέρουμε ότι θέλουν ε, οπωσδήποτε όταν πρόκειται για Αμερικανούς πολίτες να τους διαβιβάζονται τα στοιχεία στις Ηνωμένε Πολιτείες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στα συνδέει όλα αυτά στις προτάσεις που καταθέτει, δηλαδή να υπάρχει μια αμοιβαιότητα και οι Ηνωμένε Πολιτείε να δίνουν και σε εμά φορολογικά στοιχεία για τους δικούς μας πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφα. Και τώρα θα περάσουμε στην Επιτροπή ΕΚΟΝ. Πρώτος ο κύριος Νίτερ Μάιερ, ο συζητητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Χαίρομαι που μπορούμε να σας βλέπουμε εδώ τελικά ασχολούμαστε με πολύ σημαντικό θέμα, κάτι την άποψή μου. Δεν ασχολούμαστε με το θέμα του ανταγωνισμού του φορολογικού, αλλά κάτι και τη διαφορά μεταξύ οικονομικής δραστηριότητα και φορολόγησης, που είναι σοβαρότατο πρόβλημα. Και υπάρχει συνένεση ότι δεν θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η πρακτική. Πρέπει να βρούμε όμως πώς να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αποτελεσματικά. Καταρχάς, σας ευχαριστώ για το έργο που επιτελέσατε μέχρι τώρα. Συμφωνούμε όλοι ότι είναι απλώς η αρχή. Μπορώ να επαναλάβω και το ερώτημα που ετέθη μόλις τώρα. Δηλαδή για τις φορολογικές αποφάσεις tax, τύπου tax ruling. Ξέρω ότι αυτές οι αποφάσεις είναι μόνο ένα κομμάτι του προβλήματος. Είναι πολύ πιο περίπλοκο το γενικότερο θέμα και όλα τα συναφή προβλήματα και θα πρέπει να βασιστούμε ίσως εν μέρη και στην ανάλυση του ΟΣΑ όσον αφορά τις τεχνικές. Τεχνικές μέσω των επιχειρήσεων μετακινούν τις φορολογίες, τη φορολογία από χώρα σε χώρα για να πληρώνουν χαμηλότερο φόρο. Θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτές τις πληροφορίες. Τώρα έχω γενικές ερωτήσεις, γιατί μόλις ξεκινούν οι εργασίες μας. Η πρώτη μου ερώτηση. Ποια μέτρα προσωπικά θεωρείτε ότι είναι τα καλύτερα, ότι υπόσχονται περισσότερα στο πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το θέμα. Αυτά τα μέτρα Πώς θα εξασφαλίσουν ότι θα επιφέρουν βελτιώσεις και σε ένα λογικό κόστος. Ελπίζω ότι οι πολιτικές θα εδράζονται επί Άρα θα γνωρίζουμε επακριβώς τους στόχους μας, τους στόχους των πολιτικών και θα ξέρουμε και ποια θα είναι τα αποτελέσματα και συνέπειες. Δεύτερο ερώτημα. Πώς βλέπετε το ρόλο της διαφάνειας και των καθορισμών προτύπων στην όλη προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής όσον αφορά τη φορολόγηση των εταιριών. Ποια μέτρα μπορούν να βασίζονται στη διαφάνεια και στον καθορισμό προτύπων. Αντίστροφα, σε ποιους τομείς θεωρείτε ότι χρειάζεται κάποια νομοθετική πρόταση ή προτάσεις, διότι η διαφάνεια ή τα πρότυπα από μόνα τους δεν νομίζω ότι αρκούν. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή τύχη με τις εργασίες σας στον τομέα. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Άλλος συνηγητής της Οικονομικής Επιτροπής είναι η Αναλής Λότς. Καλησπέρα. Καταρχάς απευθυνόμενοι προς τον Επίτροπο, καλωσορίζω τα όσα είπατε και τη γενική σας προσέγγιση στον αφορά το θέμα. Ήταν άκουσα ενθαρρυντικά αυτά που άκουσα η αφοσίωσή σα στην φορολογική δικαιοσύνη είναι απτή. Έχω σύντομε τρει ερωτήσει όπω και άλλοι πολιτικοί που είχαν τρει ερωτήσει. Πρώτα απ' όλα, σχετικά με τη διαφάνεια και την καταχώρα υποβολή εκθέσεων. Θα συμφωνείτε ότι γίνεται προσπάθεια να εισαχθεί αυτό στα πλαίσια της οδηγίας για τα δικαιώματα των μετόχων. Και αυτή είναι μια προσπάθεια που στηρίζω, διότι ήδη υπάρχουν σημαντικά στοιχεία ότι εν συγκρίση με άλλου τομεί αυτό θα μας βοηθούσε να έχουμε πληροφορίες, ούτως ώστε οι επενδυτές. Ε, λοιπόν, η PwC ε, πρότεινε ότι κατά χώρα υποβολή εκθέσεων μπορεί να βελτιώσει ανταγωνιστικότητα, να αυξήσει την δανειοδότηση και να αυξήσει την χρηματοστική σταθερότητα. Και οι πρόεδροι και οι διοικητές διαφόρων επιχειρήσεων θεωρούν 6 στους 10 ότι οι πολυεθνικές θα πρέπει να απαιτείται να δημοσιεύουν τα έσοδά τους, τη φορολόγησή τους κατά χώρα. Λοιπόν, παροτρύνω τον Επίτροπο για το εξή. Θα ήταν δεδειγμένο να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν ταχύτερο προς αυτήν την κατεύθυνση, ότι τα στοιχεία υπάρχουν. Όμως, αν υπάρχουν απαιτήσει για περισσότερα στοιχεία, προτείνω μια πλήρη ανεξάρτητη αξιολόγηση στο βαθμό του δυνατού. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θυμάται αυτά που είπε στην ανακοίνωση ότι τα ωφέλη του CBCR θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όπως και το κόστος. Εν συντομία, καλωσορίζω αυτά που είπε ο Επίτροπος όσον αφορά το κώδικα και τη σχετική επιτροπή. Νομίζω ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε και να εξετάσουμε πώς λειτουργεί. Θεωρείται ότι η αναθεώρηση της, του Φόρουμ για την Κοινή Τιμολόγηση που εστιάστηκε στην πρόληψη της διπλής φορολόγησης και όχι πολύ στην πρόληψη της διπλής μη φορολόγησης θα πρέπει να εξεταστεί το πώς κινείται αυτή η Επιτροπή. Μετά, στην ομάδα μου θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε τελικά κοινό ορισμό των φορολογικών παραδείσων στην Ευρώπη και μαύρο κατάλογο των εταιριών που προσφεύγουν στου φορολογικού παραδείσου. Για να γίνει αυτό πρέπει να εντοπίσουμε και να καθορίσουμε τι επιβλαβεί φορολογικέ πρακτικέ. Ξέρω ότι η γαλλική κυβέρνηση ξεκίνησε ένα σύστημα τύπου ραντάρ που θα καταρτήσει κατάλογο ε, ανάρμοστων φορολογικών ε, συμπεριφορών. Μήπως αν γίνει αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους μακροπρόθεσμους στόχους μας. Ευχαριστώ συνάδελφε. Θα δώσω στον Επίτροπο το μικρόφωνο να απαντήσει σε ερωτήσεις των εισηγητών και μετά θα περάσουμε στις ερωτήσεις των μελών. Κύριε Επίτροπε. Ε, σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας. Βλέπουμε πόσο επίγει πολιτικά το θέμα αυτό και ποιο είναι ο τρόπος να το αντιμετωπίσουμε με απόλυτη αποφασιστικότητα. Χρειάζεται μια θετική αγαστή συνεργασία αγώνιμη Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι εκθορών Ουκάνευ. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι, αλλά είμαι στη διάθεσή σας να ξανάρθω αργότερα εν ευθέτω χρόνο, όποτε φρονείτε εσείς, για να δούμε πώς θα προχωρούν οι εξελίξεις και οι προτάσεις μας. Σήμερα ο θέμητος φορολογικός ανταγωνισμός είναι ε, γνωστή η πρακτική ε, είτε για τη λεγόμενη βελτιστοποίηση είτε με επιθετικούς τρόπους είναι απολύτως απαράδεκτη για τους πολίτες αυτή η πρακτική και δεν θα πρέπει να δείχνουμε ατολμία ή ε, να ολιγορούμε αλλά να προχωρήσουμε για να προωθήσουμε για την ε, ανταγωνιστικότητα. Δεν χωράει καμία αμφιβολία. Έγινε και μια ερώτηση τώρα για το πώς συνεργαζόμαστε με τον ΩΣΑ. Θέλω να καλωσορίσω ε, την ε, πρωτοβουλία BEPS για τη διάβρωση της βάσης και τη μεταφορά των κερδών. Είναι μια ρηξικέλευτη πρωτοβουλία και το ίδιο το G20 προχώρησε και εγώ με την προηγούμενη ιδιότητα, με τον ε, Βρετανό, Γερμανό, Ιταλό, Ισπανό ομολογό μου, θελήσαμε από την αρχή στο πλευρό του Άγχελ Χουρία να ε, βοηθήσουμε και πραγματικά ήταν πολύ έντονη επιθυμία και από πλευράς του ΩΣΑ. Υποστηρίζουμε τον ΩΣΑ, έχουμε αναλάβει κάποιες ε, δεσμεύσεις και τις προωθούμε και αυτές. Θα ήθελα όμως να πω ταυτόχρονα το εξή. Το σχέδιο του ΩΣΑ, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, είναι ακόμα υποσυζήτηση. Δηλαδή, να υπάρχει ένα αυθόρμητο εθελούσιο σύστημα ανταλλαγής προφοριών για τα tax rulings, και για τα κίνητρα και τα πλεονεκτήματα που δίδονται. Αυτό που εμείς προτείνουμε είναι ευρύτερη ανταλλαγή απόψεων. Γι' αυτό χαίρομαι και είμαι περήφανος που η Ευρωπαϊκή Ένωση και αύριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θελήσουν να προχωρήσουν περισσότερο. Διότι, επαναλαμβάνω, πρόκειται για αυτόματη, όχι για επιλεκτική. Θα αφορά τις διασυνοριακές επίσης ε, συμφωνίες, rulings και νομικά θα είναι δεσμευτικό το σύστημα σε σχέση με τον ΩΣΑ. Καλά, ΩΣΑ έχει ένα παγκόσμιο ρόλο, είναι συντονιστικό όργανο και στη συνέχεια προχωρούν σε πολιτική ε, δέσμευση. Εμείς είμαστε κάτι παραπάνω, είμαστε ένωση με νομοθετικές αρμοδιότητες. Ο πρόεδρος Γιούνκερ ε, ήδη πρότεινε στους ηγέτες του G20 αυτή η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών να γίνεται παγκοσμίως το έκανε αυτό στο Brisbane και εγώ στο G20 στην Κωνσταντινούπολη που είναι από λίγε μέρες και θα το επαναλάβω στην Ουάσιγκτον σε λίγες εβδομάδες. Γιατί σε τελική ανάλυση γιατί να μην αισθανόμαστε υπερήφανοι αν μπορούμε να είμαστε πρωτοπόροι εμείς σε αυτή την προσπάθεια. Κάποιος αναφέρθηκε στη ΦΑΤΚΑ, ε, ο κύριος Στόιρερ, αυτή την πράξη φορολογικής συμμόρφωσης ξένων λογαριασμών. Ε, είναι αμερικανική η πρωτοβουλία για την κατάργηση του τραπεζικού απορρίτου. Και εγώ θα χαιρόμουν και θα προτιμούσα ε, για τα tax rulings τώρα να είναι ευρωπαϊκή η πρωτοβουλία και να ε, μας ακολουθήσουν οι άλλες χώρες του ΩΣΑ. Έχουμε ένα δικό μας φιλοπορίες και τον Ιούνιο θα πρέπει να είμαστε συνεκτικοί και σύμφωνοι και συνεπείς με τις συνθήκες να προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα σε στενή συνεργασία και πάλι με τον Όσα ο καθένας με το δικό του διακριτό θεσμικό ρόλο και τις μεθόδους του. Αλλά με την βούληση πάντα να βοηθήσουμε. Για τις συστάσεις αναχώρα με ρωτήσατε. Για την Πορτογαλία αύριο ε, θα μεταβώ εκεί να συζητήσουμε αυτά και άλλα θέματα μπορώ να καταλάβω ότι μια χώρα θέλει να προσελκύσει εταιρείε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι καταδικαστές όλες οι συμφωνίες rulings. Η αρχή ε, δεν είναι καταδικαστέα. Γιατί μια εταιρεία όταν επενδύει μπορεί να έχει έτσι, μια δυνατότητα να προγραμματίζει και να σχεδιάζει τι φόρους θα πληρώσει και πού. Εγώ άλλο λέω, να μην υπάρχει αυτή ή ε, συγκατάβαση προς εταιρείε που το εκμεταλλεύονται αυτό το ιδιαίτερα ε, ευνοϊκό σχήμα ε, και να το γνωρίζει μια χώρα αυτό εις βάρος των άλλων μελών και ερήμην τους. Βεβαίως θα πρέπει αυτά όλα να τα δούμε πιο συντονισμένα και μέσω του δικού μας πρίσματος. Αυτό κουμπώνει πάρα πολύ ωραία με την πρώτη ερώτηση του κυρίου Τόιρερ τώρα. Για ποιο λόγο και πώς θα πρέπει να λειτουργεί το δικό μας σύστημα. Γιατί αναμένω εγώ τόσο σπουδαία αποτελέσματα. Σήμερα οι ισχύοντες κανόνες έχουν πολλά παραθυράκια. Αφήνουν μεγάλο περιθώριο λιγμών στα κράτη-μέλη και έχουν και πολλές γκρίζε ζώνες. Το είπα προηγουμένως έτσι κάπως ε, γρήγορα, το ξαναλέω. Μπορεί ένα κράτος μέλος να αρνηθεί να διαβιβάσει πληροφορίες εν ονόματι του εμπορικού απορρίτου και για λόγους δημόσιας πολιτικής. Έχει τη δυνατότητα να το πράξει σήμερα και να επιλέγει ποιες πληροφορίες θα διαβιβάσει και ποιες όχι. Άρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που δεν μπορεί ε, κανείς να λάβει τις απαντήσεις που θέλει, είτε ποτέ, είτε να είναι μη πλήρης και τα λοιπά. Είναι στη διακριτική ευκαιρία εκείνους που, που κατέχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που υποτίθεται ότι τα κράτη-μέλη διαβιβάζουν το ένα στο άλλο. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας να εκτιμήσουμε ε, ποια είναι η παράβαση που θα πρέπει να ε, διώξουμε, ας πούμε, να προσφύγουμε. Μέχρι σήμερα κανένα κράτος μέλος δεν έχει προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, διαμαρτυρώμενο ότι δεν μου δίνουν πληροφορίες σε άλλα κράτη. Γι' αυτό εμείς δεν λέμε αυθόρμητη ανταλλαγή και θελούσια, αλλά αυτόματη και νομικά δεσμευτική, έτσι ώστε να υπάρξουν πολύ σαφείς απαιτήσει για το ποιες είναι οι πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζονται και με ένα αριθμό που γνωρίζετε, ανατρίμηνο. Επίσης, καταργήσαμε κάθε δυνατότητα των κρατών μελών να μειώνουν ή να αρνούνται Πλήθο ε, το πλήθος των προφοριών που θα δίνουν. Και λέω εμπαρόδο στο Κοινοβούλιο και για τα κράτη-μέλη είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει πρόσβαση σε όλες τις στατιστικές για τα στοιχεία που διαβιβάζονται και ανταλλάσσονται. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν τα κράτη-μέλη εξορισμού, αλλά νομίζω ότι αυτό το σημείο θα πρέπει εμείς και εσείς να το υπερασπιστούμε. Γιατί μπορεί κάποιος να μπει στον πειρασμό να πει Ας εξαιρέσουμε τώρα, παραγωνίσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα τα κανονίσουμε μεταξύ μας τα κράτη-μέλη. Μα σε περίπτωση που υπάρχει βαριά παράβαση θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι παρούσα. Είναι χρήσιμο αυτό. Δεν το κάνουμε για τον εαυτό μας, αλλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κύριε Τόιρερ, ε, πώς θα περάσει. Ε, δεν θα είναι ο νόμος του Γκρέσαν που λέγεται, αλλά ε, οι καλές πρακτικές θα παραγωνίσουν τις κακές. Δηλαδή θα αναγκαστούν τα κρατημέλη να υποχωρήσουν κάπως ε, από αυτή την ε, υπερβολική εύνοια και επίσης οι επιχειρήσεις θα το δουν ως αντικίνητρο αυτό. Η κοινή γνώμη, έστω και ε, σιωπηρά, είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγον γιατί η δικαιοσύνη γεννιέται μέσα από τη διαφάνεια. Άρα θα το γνωρίζουν και οι εταιρείε αυτό. Και θα έχει αποτέλεσμα για τον κανόνα, μάλλον τον κώδικα συμπεριφορά και διοντολογία. Στο παρελθόν λειτουργήσε. Εντάξει. Οι μέθοδοι και οι δυνατότητες διερεύνησης πλέον που παρέχει δεν είναι στο επίπεδο της εξειδίκευσης ε, της περιπλοκότητας που χρησιμοποιούν για τα tax rulings οι εταιρείε και οι χώρες. Αλλά ε, δεν είναι υποκατάστατο ε, αυτό που προτείνουμε, είναι νομοθετικό μέσο. Για τους Υπουργούς Οικονομικών βεβαίως θα τους προτείνω κατά τη διάρκεια των διμερών μας επαφών να έρχονται πιο συχνά, αλλά αυτό που έχει σημασία και για την Επιτροπή Τάξη και για την Επιτροπή ΕΚΟΝ είναι ότι θα πρέπει να σεβόμαστε όλοι τους κανόνες. Αν το εγχείρημα εδώ στο Κοινοβούλιο είναι, παραμείνει ατελές, δεν θα έχει νόημα, δεν θα έχει αποτέλεσμα και δεν θα πείσει κιόλα. Θα πρέπει ε, οι πάντες να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τη δική σας Επιτροπή και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν έχει τίποτα να κρύψει, για τα κράτη-μέλη που κανονικά δεν θα πρέπει να έχουν τίποτα να κρύψουν. Και ελπίζω και οι Υπουργοί Οικονομικών να εφορούνται από το ίδιο πνεύμα. Για τη ΦΑΤΚΑ, την πράξη φορολογικής συμμόρφωσης ξένων λογαριασμών, ε, ξέρετε το 2016 θα έχουμε παγκόσμια πρότυπα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, η αρχή της αμοιβαιότητας, στην οποία αναφερθήκατε. Κύριε Νίντερ Μάιερ, με ρωτήσατε για τα πιο ε, φερελπίδα μέτρα για το μέλλον. η διαφάνεια, η πίεση των μοτίμων, αυτό το peer pressure, για να προχωρήσουμε όσο γίνεται περισσότερο, αλλά για την εσωτερική αγορά αυτό που έχει σημασία είναι να καταλήξουμε στο CCCTB που είναι κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιριών. Από το 11 ε, που άρχισε αυτή η προσπάθεια έχουν περάσει 4 χρόνια. Μπορούμε είτε να πάρουμε τις ε, ίδιες προτάσεις και να τις εγκρίνουμε αλλά το πρόβλημα είναι ότι τα ίδια αίτια οδηγούν στα ίδια αποτελέσματα. Μπορεί να θεωρήσουμε ότι έχουν οριμάσει κάπως περισσότερο τα κράτη-μέλη. Μπορούμε και αυτό να το τσεκάρουμε. Ή να αλλάξουμε τακτική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποκλείει τίποτα από όλα αυτά. Τα επεξεργάζεται. Και μετά υπάρχει και ενισχυμένη συνεργασία που είναι η έσχατη λύση γιατί αυτό αποδεικνύει ότι αν δεν μπορείς να προχωρήσεις ε, με τους 28 πασαλού, αλλά θα πρέπει και οι 28 να συνεργαστούν. Στο πρόγραμμα δράση λοιπόν που εμείς και εγώ προσωπικά προετοιμάζουμε και εκπονούμε, θα συμπεριλαμβάνω είναι πάρα πολύ σημαντικά. Για την κυρία Ντότς. Το ταχύτερο δυνατόν θα γίνει εξολόγηση συνεπιών, ούτω ώστε να ετοιμαστεί. Ανεξάρτητη μελέτη είναι κάτι Είναι καλή ιδέα, καλύτερη ιδέα διότι πρέπει να πετύχουμε πλήρη διαφάνεια και πλήρη αξιοπιστία στα μέτρα μας. Και βέβαια η ανεξαρτησία είναι βάση για αξιοπιστία και διαφάνεια. Κοινό βήμα το φόρουμ για την κοινή τιμολόγηση. Καλώς θα δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί η λειτουργία αυτού του φορέα. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα επανέλθουμε τώρα σε ερωτήσεις των μελών. Η κυρία Ντανούτα Ήμπνερ είναι πρώτη εν ονόματι του ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Έχω δύο ερωτήσεις. Η μία σχετίζεται με την έρευνα που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά των τεσσάρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η νομική βάση είναι το 107, άρθρο 107 για τις κρατικές ενισχύσεις. Έχουμε και το άρθρο 116. Γνωρίζουμε ότι δεν αφορά μόνο το θέμα κρατικών ενισχύσεων αλλά σε καποια κάτι κράτη-μέλη αφορά και δράσεις, όχι μόνο διατάξεις. Δράσεις διοικητικής φύσεως που οδηγούν σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού της εσωτερικής αγοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει και την άλλη νομική βάση στην όλη προσπάθειά της για το μέλλον. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Συζητούμε τον φόρο των επιχειρήσεων, αλλά έχουμε και τον φόρο προστιθέμενης αξίας και, οποιος, και οποιοδήποτε φορολογούμενος που θέλει να κάνει διασυνοριακή συναλλαγή μπορεί να ζητήσει απόφαση σχετικά με το ΦΠΑ, ruling δηλαδή, και να τη λάβει. Η ερώτησή μου είναι, ξεκίνησε δράση εδώ και αρκετά χρόνια μια δράση και έγινε κάποιο πιλωτικό πρόγραμμα. Εξέταζε τις συμφωνήσεις ιδιωτικές, τα rulings για το ΦΠΑ. Συνεχίζει προσπάθειες Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ντανούτα. Για τους σοσιαλιστές, ο, κύριο κύριος Πίτερ Ζήμεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να συνεχίσω από αυτά που, που είχα πει την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλεια. Δύο ερωτήματα για τη διαφάνεια. Είπατε ε, πώς είχε η κατάσταση, το είπε και ο κύριος Τόιρερ, ορισμένες υποχρεώσεις του παρελθόντος δεν ε, ε, υλοποιήθηκαν. Ερώτηση συγκεκριμένη στο μέλλον. Σκέφτεστε και τίποτα κυρώσεις ή θα είναι μόνο υποχρέωση που θα γράφεται με πιο έντονο και πιο οξύ τρόπο ή εάν τα κράτη-μέλη δεν το τηρήσουν όλα αυτά, τι θα γίνει, θα προβλέπονται και κυρώσεις. Δεύτερη ερώτηση και αφορά τα κεντρικά μητρώα για τα tax rulings. Εδώ για το ξέπλυμα χρήματος, την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έχουμε διάφορες μορφές μητρών. Ε, είχε γίνει μεγάλος καυγάς Κοινοβουλίου, Συμβουλίου τότε. Θα είχε μεγάλο νόημα να υπάρχουν τέτοια μητρώα ε, και να είναι και δημόσια. Βέβαια δεν θέλω να μπω στο φορολογικό απόρριτο και σε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά τα βασικά στοιχεία ε, θα μπορεί να είναι χρήσιμα για το κοινό και να βλέπει ο καθένας ποιος πληρώνει τους φόρους του σε ποιο κράτος. Και ε, στη συνέχεια, υπάρχουν κάποιοι που είναι σύμβουλοι μεγάλες διεθνείς εταιρείες και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών και των εταιριών είναι και μεγάλα διεθνή δικηγορικά γραφεία. Ε, Ασχοληθήκαμε και για τους σημαίνους οίκους αξιολόγησης και με κάποια μεγάλα γραφεία λογιστικού ελέγχου τι γίνεται με τη σύγκρουση συμφερόντων και τη διαπλοκή. Για το συγκεκριμένο δεν βλέπω καμία πρόταση. Προτίθεται να το κοιτάξει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενδιαφέρει και την Επιτροπή ΤΑΞ. Ε, θα κοιτάξετε και που υπήρξαν ε, στο παρελθόν τέτοιες συγκρούσεις συμφερόντων, σε ποιο βαθμό και σε ποια ένταση αν υπήρχαν αυτές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ εν ονόματι του ECR, ο κύριος Μπεντ Λούκε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρο. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε που ήρθατε σήμερα στην ακρόαση εδώ για να μας απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. Καταρχάς πρέπει να πω ότι θεωρώ πολύ καλή καταρχήν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την πρωτοβουλία αυτή. Υπάρχουν όμως και ανοιχτά ερωτηματικά και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά. Πρώτον, μιλήσατε για την μελέτη επιπτώσεων. Γιατί θα το κάνετε αυτό για το μέλλον. Δεν μπορείτε να αξιολογήσετε εκ των προτέρων ε, αυτά που θέλετε να προτείνετε, τι επιπτώσεις θα έχουν. Πώς θα επηρεάσει τη φορολογική διοίκηση κάθε κράτους αυτό που προτείνετε. Η φορολογία, δηλαδή η εφορία κάθε τρεις μήνες θα παίρνει από τα 28 κράτη-μέλη στοιχεία και θα πρέπει να τα ελέγχει δεν σας πιστεύω πάρα πολύ ότι αυτό δεν σημαίνει τεράστιο κόστος ε, διοικητικό για την εφορία της κάθε χώρας. Και θα ήθελα ε, να μάθω και την άποψη της εκάστοτε εθνικής φορολογικής αρχής. Αυτό είναι ε, και το αντολαμβάνονται αυτοί ως ένα μέτρο καταπολέμησης της γραφειοκρατίας ή ως τεράστιο φόρτο εργασίας επιπλέον που θα τους κατακλείσει. Δεύτερη ερώτηση. Είπατε ότι οι ε, φορολογούμενες εταιρείες έψαχναν ε, μανιωδώς φορολογικά πλεονεκτήματα. Αυτό μπορεί να ισχύει για κάποιες εταιρείες, αλλά υπάρχουν και άλλες εταιρείες που δεν ε, ψάχνουν με μανία αυτές τις ρυθμίσεις, αλλά έρχονται με μανία κάποιες εφορίες και τους χτυπάνε την πόρτα και με προτάσεις και προσφορές για το πώς μπορείς να πληρώσεις τους λιγότερους φόρους. Δηλαδή η τεχνική της φοροαποφυγής είναι να δούνε και λαβήν. Δεν είναι μόνο οι εταιρείε που ψάχνουν, ψάχνουν και οι εφορίες και μάλιστα αγρίως. Οπότε με τη διαφάνεια και μόνο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την εκατέρωθεν επιθυμία φοροαποφυγής και αν οι ε, εφορίες υποχρεώνονται να δημοσιεύουν τα επίσημα στοιχεία, ποιος μας εγγυάται ότι δεν υπάρχουν παράλληλες υπόγειες διαδρομές που είναι τελείως διαφορετικές από το φορολογικό σημείωμα και το εκαθαριστικό το οποίο δημοσιεύεται. Και πώς θα εξασφαλίσετε εσείς ότι δεν θα γίνεται αυτό το ruling όπως γίνεται και σήμερα, απλώς υπογείως και θα δημοσιεύονται άλλα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κόρα Βανιούεν Όιτσεν, Αξονόματος του Άλντε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, εδώ είμαι πίσω, πίσω. Καλώς ήρθατε ξανά κύριε Μοσκοβίτση. Χαίρομαι που ξαναβλέπω τόσο σύντομα. Συζητήσαμε και την περασμένη εβδομάδα και στην Ολομέλεια. Στην Ολομέλεια λοιπόν όπως σας είπαμε τότε, καλωσορίζει Άλτε την, πρωτο, την πρωτοβουλία σας για την οδηγία για διαφάνεια φορολογική. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, οι εθνικές φορολογικές αρχές να αναφέρουν κάθε διασυνοριακές συμφωνίες rulings που έχουν εκδοθεί. Όλα τα κράτη-μέλη. Δεν θα ήταν αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο αν τα κράτη-μέλη ανταλλάσσουν πληροφορίε μόνο με εκείνα τα κράτη-μέλη τα οποία ενδεχομένω εμπλέκονται με τη φορολογική δομή τη σχετική επιχειρήσεω αντί να μοιράζονται όλες τις πληροφορίες με όλους. Δεν θα έπρεπε να εστιαστείτε στις συγκεκριμένες πληροφορίες. Ήταν η πρώτη ερώτηση. δεύτερη ερώτηση. Οι απαιτήσει ποιότητα των αφορά πληροφορίε που θα ανταλλάσσονται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώ θα υποπτεύει και θα επιβάλλει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των συναλλασσομένων πληροφοριών. Διότι ένα ruling μπορεί να είναι ruling, αλλά μπορεί να υπάρχει μια συμφωνία που να είναι τύπου ruling, αλλά να μην αναφέρεται. Όπως είπε ο κ. Λούκε, θα έπρεπε ίσως να λάβουμε υπόψη και πράγματα τα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί επισήμως ως ruling, αλλά μπορεί να εμπεριέχουν σημαντικές πληροφορίες. Μπορεί, πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε την ποιότητα των πληροφοριών. Τελική ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι θα αξιολογήσει τις συνέπειες δημόσια αποκάλυψης άλλων πληροφοριών στον αφορά τη φορολόγηση των εταιριών πέραν τις πληροφορίες για τα συμφωνίες τύπου rulings. Σε ποιες πληροφορίες αναφέρεστε? Πώς θα αξιολογήσετε τον αντίκτυπο ενδεχόμενης αποκάλυψης άλλων πληροφοριών, πώς θα γίνει αυτή η αξιολόγηση των συνεπειών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κόρα. Για την ΚΟΕ, ο κύριος Φάμπιο Ντεμάση έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Μοσκοβησή. Στη ε, φορολόγηση των επιχειρήσεων ε, έχουμε νόμιμο φορολογικό dumping που είναι αθέμητο και οργανωμένη ε, εγκληματικότητα με μεγάλη υποστήριξη και οικονομικών και υπουργών οικονομικών. Και ο κύριος Γιούγκερ τα γνωρίζει αυτά και θα ήθελα να τονίσω εξ ονόματος της Επιτροπής μου, της ομάδας μου, συγγνώμη, ε, ότι ενθαρρύνουμε whistleblowers, ανθρώπους να καταγγείλουν ε, πράγματα που γνωρίζουν, όπως ε, φαίνεται από τη διερευνητική δημοσιογραφία και τον Guardian, από στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας. Από το 1977 υπάρχουν συστήματα ε, εθελούσιας ανταλλαγής προφοριών 38 χρόνια τώρα και εγώ είμαι 35 ετών, δηλαδή πριν γεννηθώ. Γέννητος ήμουνα όταν τα ρυθμίσατε αυτά και είναι αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεματοφύλακας των συνθηκών να εξασφαλίζει και να παρακολουθεί αυτές τις ανταλλαγές. Γιατί εξ όσων γνωρίζω οι οδηγίες παραμένουν οδηγίες, δηλαδή κοινοτικό δίκαιο. Ανεξαρτήτως της οξύτητας ε, ε, της διατύπωσης εν και κείμενη νομοθεσία σημαίνει ισχύον δίκαιο. Τι έχει κάνει στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί το 2011 την αναθεωρήσατε αυτή την οδηγία. Και το δεύτερο είναι ότι εγώ δεν εμπιστεύομαι ε, τους Υπουργούς Οικονομικών. Ξέρουμε τη συζήτηση για τη λίστα Λαγκάρτ που είχε η προηγούμενη ελληνική κυβέρνηση στα χέρια της και σε τι ε, οδήγησε. Και θέλω να ρωτήσω και σε σχέση με τα όσα είπε ο Πέτερ Ζήμων. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να είναι ε, δημόσια σε ενδιαφερομένους ειδικού από την κοινή γνώμη, γιατί εγώ δεν εμπιστεύομαι απλούστατα τους υπουργού Οικονομικών ότι δεν θα τα βάλουν σε ένα σερτάρι για να ξεχαστούν. Εσείς από πού αντλείτε αυτή την εμπιστοσύνη. Επίσης, θα ήθελα να γνωρίσω εάν έχετε μάθει τα όσα έκανε η ε, εταιρεία Χρυσού Ελντοράντο στα Κανάρια ε, με... Ε, συγγνώμη, από, τον Καναδά, το Ελντοράντο, σε σχέση και με την ελληνική κυβέρνηση, η εταιρεία Χρυσού έχει συνεργαστεί και με Ολλανδούς και ε, ε, μάλιστα ο Ολλανδός, ο Υπουργός Οικονομικών εμποδίζει αυτή τη στιγμή την Ελλάδα ε, να καταβάλει το χρέος της όπως η ίδια επιθυμεί και έχει δεσμευτεί. Τι θα κάνετε λοιπόν, θα κάνετε κανένα διάβημα προς τον κύριο Ντάισελμπλουμ και αν δεν έχετε τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται σήμερα για την καναδική εταιρεία να σας τα δώσω, τα έχω φέρει. Και επίσης οι τράπεζες βοηθούν ε, τις επιχειρήσεις να φοροδιαφεύγουν σε διάφορους φορολογικούς παραδείσους γιατί έχουν εκεί τις ιατρικές και υποκαταστήματα. Ε, προτίθεστε να προβείτε σε καμία κύρωση εναντίον των τραπεζών αυτό να τους αφαιρέσετε την άδεια λειτουργία στην Ένωση ας πούμε. Ευχαριστώ μόλις κάτω για τους πρασίνους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Ευπρόσδεκτα τα αρχικά σας σχόλια και η δέσμευσή σα για κατεπίγουσα και σοβαρή πρόοδο για να αποφευθεί η φοροαποφυγή. Και συμμερίζουμε την άποψή σα, Έχουμε ιδιαίτερο ρόλο να διαδραματίσουμε με μια ενιαία και πλούσια αγορά. Να καθορίσουμε διεθνεί προδιαγραφέ για του κανονισμού περί φορολογήσεω εταιριών. Αν θέλουμε να πετύχουμε του στόχου μα, δεν θέλουμε να έχουμε τόσο μελέτε και εκθέσει και διαφάνεια, θέλουμε να ακούσουμε περισσότερα για κανόνε, πρόστιμα και επιβολή. Επίση, η εμπιστοσύνη μας στην προθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δράσει υπονομεύεται από κάποιες πτυχές του περασμένου ιστορικού και της απροθυμίας προηγούμενων επιτρόπων να κινηθούν όταν είχαν σαφή στοιχεία παραβιάσεως των υφισταμένων ε, νόμων που ήδη αναφέρατε. Παράδειγμα, διαπιστώσαμε ότι στις 17 Απριλίου του 2012 στον Εντογικό Κώδικα, στην ομάδα του Εντογικού Κώδικα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε απογοήτευση των αποτελέσματα της ερωτήσεων που έβαλε σε κράτη-μέλη στον αφορά ανταλλαγή πληροφοριών. Το Βέλγιο τότε πήρε το λόγο και δήλωσε ότι δεν είχε ανταλλάξει εσδήποτε πληροφορίε διότι δεν είχε λάβει καμία πληροφορία από άλλα Αργότερα το Συμβούλιο, νομική υπηρεσία του Συμβουλίου, διευκρίνησε την κατάσταση και είπε ότι δεν υπήρχε νομική υποχρέωση για αμοιβαιότητα όσον αφορά την οδηγία περί διοικητική συνεργασία ή για την προηγούμενη ε, οδηγία περί αμοιβαία αρρωγή. Οπότε υπήρχαν σαφή στοιχεία παραβάσεω, αλλά δεν υπήρχαν αντίστοιχα στοιχεία δράσεω που ανελήφθη, ούτω ώστε να επιβληθούν υποχρεώσει που υπήρχαν τα κρατημένα να συμμορφωθούν με τον κώδικα. Σε αυτή την υπόθεση, όπω ανέφερα, το Βέλγιο είχε απράξει το δίκημα αλλά είδαμε από τη συνεδρίαση, είπε το Βέλγιο ότι και άλλα κράτη-μέλη δεν είχαν πληρώσει προχρεώσει του. Τι υπονοούσε ότι η Ιρλανδία δεν ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την απόφασή τη για, το για την Apple και το Λουξεμβούργο για την απόφαση περί Amazon. Δεν ενημέρωσε άλλα κράτη-μέλη. Τα γνωρίζουμε αυτά. Γνωρίζουμε επίση, όπω είπε και συνάδελφο Φάμπιο, ότι αυτή η υποχρέωση υπήρχε από τη δεκαετία του 70 και τα κράτη-μέλη υπήρχαν υποχρέωση ανταλλαγή πληροφοριών περί των συμφωνιών των φορολογικών rulings έκτοτε. Η ερώτησή μου, πρώτον, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μην ξεκινήσει η διαδικασία κατά παράβαση όταν δέχτηκε το Βέλγιο ότι δεν συμμορφώθηκε υποχρεώσει σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και υπενόησε ότι και άλλα κράτη-μέλη δεν αντάλλαξαν πληροφορίε. Δεύτερον, Είσαστε έτοιμο να δώσετε οδηγία στι υπηρεσίε σε αυτή τη φάση να γίνουν τα πρώτα βήματα προ διαδικασίε κατά παράβαση. Νομίζω ότι τέτοια δράση επιβολή ενδείκνυται. Θα ήταν σημαντικό βήμα να δείξει ότι είναι σοβαρή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την αντιμετώπιση τη ε, φοροαποφυγή από τι επιχειρήσει και των συμφωνιών φορολόγηση tax rulings. Ευχαριστώ πολύ. Εν ονόματι του ευτή, ο κύριος Μάρκο Τζένι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εσείς είπατε ότι το πακέτο για τη διαφάνεια είναι απλώς ένα πρώτο βήμα και δεν αρκεί. Εγώ προσθέτω ότι κατά την άποψή μου δεν είναι κατελάχιστον αρκετό για να αντιταχθεί σε αυτή την επέσχυντη δραστηριότητα. Εγώ ντρέπομαι που σκέφτομαι ότι μετά από περίπου 25 χρόνια από την υπογραφή της συνθήκης του Μάστρικτ είμαστε εδώ και συζητούμε ακόμα αυτά τα προβλήματα όταν κάνουμε, βγάζουμε διάφορους λόγους για την ενιαία αγορά, για την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, βλέποντας την τεράστια πίεση που ασκούν τα μέσα που οδήγησε η πίεση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, εγώ περίμενα μια πολύ πιο γενναία ε, προσέγγιση από την αρχή. Από το πρωί φαίνεται η καλή μέρα. Εγώ δεν περιμένω τίποτα πολύ καλό ούτε από το πακέτο του Ιουνίου, αλλά ελπίζω να κάνω λάθος. Όσον αφορά τη διαφάνεια, κάτι θεμελιώδες, είναι καλή η διαφάνεια, αλλά είναι καλό η διαφάνεια να δούμε ότι αυτή καθ' αυτή δεν οδηγεί σε φορολογική δικαιοσύνη. Και αυτό θα πρέπει να είναι τελικά ο στόχος. Θα πρέπει να εστιαστούμε επί του πραγματικού προβλήματος και να προσπαθήσουμε να εξεύρουμε λύσεις επ' αυτό. Όσον αφορά το πακέτο για τη διαφάνεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις από εσά, διότι κατά την άποψή μου δεν υπάρχει αρκετή σαφήνεια. Πρώτα σε μια απάντηση είπατε ότι η κοινή γνώμη είναι ένα θεμελιώδες ε, στοιχείο για τη διαφάνεια. Όμως θα ήθελα να γνωρίζω γιατί στο πρώτο πακέτο για τη διαφάνεια που παρουσιάσατε αυτές οι ανταλλαγές των πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών δεν θα είναι δημόσιες, δεν θα αποκαλύπτουν στο δημόσιο, στο κοινό. Διότι για σας αυτό το στοιχείο είπατε ότι είναι θεμελιώδες. Ένα άλλο σημείο για το οποίο δεν διέπεται, δεν υπάρχει ένα πλαίσιο για την αλλαγή πληροφοριών. Τα ανέφερε άρθρο στην Τεμάτζη. Τίποτα δεν εξασφαλίζει ότι πραγματικά υπάρχει βούληση από πλευρά των Υπουργών Οικονομικών να ανταλλάξουν αυτέ τι πληροφορίε. Και κάτι άλλο, όσον αφορά τη δουλειά που θα πρέπει να κάνει η Επιτροπή, η Γενική Διεύθυνση, η Γενική Διευθύνση τη Επιτροπή για να αντιμετωπίσουν τον όγκο αυτών των πληροφοριών. 22 από τι 28 χώρε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω εφαρμόζουν αυτά τα tax rulings. Αυτό σημαίνει ότι θα φτάσει ένας μεγάλος όγκος πληροφοριών ε, θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν σε αυτή τη φάση αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποια δομή που είναι ικανή να αντιμετωπίσει και να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά αυτό τον όγκο των πληροφοριών και αυτό το είδος των πληροφοριών. Και κάτι άλλο θεμελιώδες είναι η χρήση των Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων. Εγώ θα ήθελα πραγματικά να πάρουμε σαν παράδειγμα την εμπειρία της ομάδας των εμπειρογνωμόνων όσον αφορά το transfer pricing και να θέσουμε σαν βάση αυτό για να χρησιμοποιήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Η ομάδα για το transfer pricing απαρτίζεται αποκλειστικά από μέλη που είχαν κάθε συμφέρον να παραμείνει η καθεστική ατάξη. Λοιπόν, στην αναθεώρηση αυτών των ομάδων εργασιών, βλέποντας ότι η κοινή γνώμη κατά την άποψή της έχει κεντρική σημασία, θα πρέπει σε αυτές τις ομάδες να υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των εμπειρογνωμόνων των διαφόρων τομέων και, και να υπάρχουν και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Τελευταίο σημείο, το οποίο θα ήθελα να θίξω και θα παρακαλούσα και θα ευχόμουν στην πρόταση του Ιουνίου να ξεπεράσουμε τα προβλήματα, να διαπιστώνουν τα προβλήματα, να προταθούν λύσεις, ούτως ώστε οι δομές και τα πλαίσια που θα χρησιμοποιηθούν για να ε, καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή, η οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται να γίνουν παράνομοι οι μέθοδοι για την ε, φοροδιαφόγη. Θέλουμε μια πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα είναι αποτελεσματική, που θα έχει πραγματικά αποτελέσματα. Λοιπόν, έχουμε και το corporate tax, base που υπάρχει, καλή, επρόσδεκτη και διαφάνεια, αλλά δεν αρκεί. Θα πρέπει να δράσουμε από αυτόν, θα πρέπει να τιμωρήσουμε τις ε, συμβουλευτικέ εταιρείε και τι τράπεζε που όπω είδαμε και όπω όλοι γνωρίζουμε βοηθούν την ε, φοροδιαφυγή. Και αυτό θα περίμενα εγώ από την πρόταση που θα υποβληθεί τον Ιούνιο και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις μία εγγεγραμμένες ο κύριος Μπερνάου Επίτροπε, η Ειδική Επιτροπή συγκροτήθηκε για να ρίξει φως σε διάφορες επιθετικές πρακτικές φοροαποφυγής και για να απευθύνει συγκεκριμένε συστάσεις καταπολέμησης αυτού του φαινομένου. Λοιπόν, βασίζομαι σε μια απλή διαπίστωση. Από το 2012 ως το 2014 είστε υπουργό Οικονομικών. Δεν μπορεί να αγνοούσατε τις ε, ε, ε, έκνομες πρακτικές του Λουξεμβούργου. Γνωρίζατε τα περί δημοσιονομικού ελλείμματος, δημοσιονομικού δημοσιονομικού που σας εκκληροδότησε ο συνάδελφός από το ΙΕΜΠ. Δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ φορολογικών εσόδων έχουν απολεστεί έτσι. Αυτό δεν σας ενοχλεί. Ε, φέρνει σε ανισορροπία τον προπολογισμό της Γαλλίας. Λοιπόν, ποια συγκεκριμένα μέτρα θα αναλάβετε ούτως ώστε να κάνετε κάτι πέρα από τις ε, δηλώσει καλή θέληση. Ε, θα πάρω δύο συγκεκριμένα παραδείγματα που προκύπτουν από εκθέσεις του Κοινοβουλίου. Πρώτον, θα περιορίσετε ή θα απαγορεύσετε τις ε, την πρόσβαση στα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, των επιχειρήσεων που εγκαθίστανται σε φορολογικούς ε, παραδείσους ή λαμβάνουν παράνομες κρατικές επιδοτήσεις. Και δεύτερον, θα κάνετε κάτι κατά των εταιριών που συμβουλεύουν, δίνουν συμβουλές για αυτήν την φορολογική βελτιστοποίηση. Για τα τελευταία χρόνια θα επιβάλλετε κυρώσεις στα κράτη-μέλη ε, ε, θα επιβάλλεται καιρό στι επιχειρήσει που έχουν ακολουθήσει την εφορολογική βελτιστοποίηση, ούτω ώστε να υπάρξει αποζημίωση των κρατών μελών. Θα υπάρξει κάλυψη των ζημιών ε, των κρατών μελών από πλευρά των επιχειρήσεων θα επιστραφούν οι φορεί, στα κράτη-μέλη όπου κανονικά θα έπρεπε να έχει επέλθει φορολόγηση. Έχει την πρόθεση να το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ποια ε, μεθοδολογία υπολογισμού θα χρησιμοποιήσει. Θα ήθελα να μου δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις. Ευχαριστούμε, λέει ο κ. Λαμασούρ. Κάναμε ένα γύρο και ακούσαμε ε, το, σε εκπροσώπους όλων των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο πρωτού περάσουμε στο δεύτερο γύρο. Ευχαριστώ. Θα αρχίσω από την αρχή, από τις ερωτήσεις ε, της κυρίας Χιούμπνερ. Συγγνώμη, δεν θα απαντήσω ε, στην πρώτη, διότι είναι αρμοδιότητα της συναδέλφου Μάγκρετ Βαστεγκέρε και εκείνη ε, μπορεί να σας απαντήσει συγκεκριμένα με δεδομένα. Εξορισμού δεν μπορώ να γνωρίζω τις απαντήσεις. Η Γενική Διεύθυνση ε, για τον Ανταγωνισμό και η Επίτροπος ε, με την προσήλωση που τους χαρακτηρίζει θα καταλήξουν σε συγκεκριμένα ε, στοιχεία και θα σας τα κοινοποιήσουμε. Δεν είναι κράτος εν κράτη, όμως θα πρέπει να σεβαστούμε το ότι πρόκειται για διαφορετικές δομές, διαφορετικές υπηρεσίες. Για το ΦΠΑ έχουμε κατοχυρώσει την διοικητική ανταλλαγή πληροφοριών και για την περίοδο 2007-2017 ο στόχος μας είναι να είναι να παγιοποιηθεί πλέον το σύστημα για το ΦΠΑ μετά από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα κατατεθεί μεταγενέστερα για να μην προκύψει ε, νομοθετική συμφόρηση ε, πάντως, κατά τη γνώμη μου, μελλοντικά τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να επιλέξουν ε, για ποια προϊόντα θα έχουν το μειωμένο συντελεστή του ΦΠΑ. Θυμηθείτε και την τελευταία απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να γίνει σεβαστή η νομολογία, όμως είναι και θέμα νομικής βάσης και στο μέλλον θα μπορέσουμε να είμαστε πιο ευέλικτοι. Για τη διοικητική ανταλλαγή των πληροφοριών για το ΦΠΑ έχουμε ήδη καταδείξει τη δέσμευσή μα. Κύριε ε, με, Μου κάνατε την ερώτηση για τις ε, κυρώσεις. Ε, αυτή η πρόταση οδηγίας ε, δεν μιλάει για ποσοτικοποιημένες εκκυρώσεις. Υπάρχει ένα στοιχείο παρόλα αυτά και επιμένω διότι Καταλαβαίνω ότι μας κάνετε ερωτήσεις ε, για το διοικητικό άχθος, ε, για τις εφορολογικές αρχές. Κύριε Λούκη, θα σας απαντήσω σε λίγο. Ε, όμως, εάν απουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν υπάρχει άλλος μηχανισμός που να οδηγεί σε ρύθμιση και άρα και επιβολή κύρωσης. Με ποια κύρωση είναι αυτή. Αν το εγγυηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, σας καλώ και πάλι να είστε σε εγρήγορση. Εάν διαπιστώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν λειτουργεί η ανταλλαγή πληροφοριών, λοιπόν τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινήσει διαδικασία επιπαράβαση και αρχίζει η διαδικασία επιβολής κυρώσεων βάσει του κείμενου μηχανισμού. Ε, με αυτόν τον τρόπο μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις. Για το Μητρό, μετά από μελέτες αντικτύπου θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες του Μητρώου. Και πάλι όμως να σας πω ότι για μένα έχει ιδιαίτερη σημασία ο πολιτικός προσανατολισμός. Κοινοποιώ, κοινοποιώ στο κοινό. Πρέπει να δούμε και ποιες επιπτώσεις θα έχει αυτό στο κοινό για τους για τις εταιρείε ε, που δίνουν συμβουλές ε, θα ήθελα να απαντήσω γιατί ακούστηκαν πολλές θετικές ερωτήσεις. Ε, για το BEPS, για τη διάβριση φορολογικής βάσης, εάν διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν ε, μετακινήσεις ε, ε, που βασίζονται σε δράσεις φορολογικών συμβούλων τμηματικά θα κινηθούμε. Για να έχουμε ρόλο πρωτεργάτη στη διαφάνεια υστερούμε λίγο στα υπόλοιπα ζητήματα προς το παρόν οπότε επίτω αυτό που λέτε και θα το εξετάσουμε στα πλαίσια αυτών που γίνονται στον ΩΣΑ αυτή τη στιγμή για μένα. Η διαφάνεια είναι κάτι που θα πρέπει να υποστηρίξουμε μέχρι τέλους και ε, για το κοινό θα πρέπει να είμαστε όσο πιο ανοιχτοί ε, γίνεται ακόμη και για τις υποχρεώσεις ε, των φορολογικών συμβούλων. Έτσι θα πρέπει να κινηθεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μην ξεχνώντας βεβαίως ότι επομίζεται τις ευθύνες της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα πρέπει να τις επομιστούν και στο Συμβούλιο και το ίδιο και η δική σας επιτροπή. Η δική σας επιτροπή θα μπορέσει επίσης να ε, χρησιμοποιήσει το βάρος της ε, σε σχέση με μελλοντικέ προτάσεις. Δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε τη σημασία του έργου σας. Ε, για την, το διοικητικό άχθος για τις φορολογικές αρχές. Ε, ε, κάθε τρεις μήνες θα υπάρχουν mails για αυτές τις φορολογικές αποφάσεις και ούτως ή άλλως υπάρχει τυποποιημένη διαδικασία για την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο στόχος είναι να έχουν τα κράτη-μέλη τα απαιτούμενα στοιχεία για να, για να υπερασπιστούν τη φορολογική τους βάση κρατώντας το ελάχιστο του φορολογικό άχθος. Λοιπόν, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να να στέλνουν ελάχιστες ε, ε, πληροφορίες υποχρεωτικά. Είναι απλούστατο το σύστημα ω προ τη συμμόρφωση. Μιλάμε για διασυνοριακή rulings, διασυνοριακές φορολογικές αποφάσεις και αυτό ε, συνεπάγεται μειωμένο διοικητικό άκθος. Δύο παρατηρήσεις όμως, εάν ε, εξετάζετε το θέμα της διαφάνειας, τότε θα πρέπει να έχετε πληρέστατες πληροφορίες ε, για να εξασφαλίσετε ότι υπάρχει διαφάνεια. Και δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα θα πρέπει η ίδια να διαθέτει αυτές τις πληροφορίες. Ο στόχος είναι να ζητούμε τα ελάχιστα αλλά και τα δέοντα. Πιστεύω θα συμφωνήσετε. Ε, για το country by country reporting σε εκθέσει κατά χώρα ε, θα αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο στην ανάλυση που έχουμε προβλέψει εξορισμού, διότι είναι, ε, δεν έχουμε τα στοιχεία στη διάθεσή μα για να κάνουμε την αποτίμηση ακριβώ επειδή είναι αδιαφανή ο τομέα. Μετά, όταν θα ασχοληθούμε με του κανόνε για την αξιολόγηση που θα συναποτελέσουν την πρότασή μα, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε περισσότερο και πάλι θα έχουμε, θα περιγράψουμε, θα ποσοτικοποιήσουμε διαφορετικές εναλλακτικέ λύσεις μετά από αντιπαραβολή και ε, έχοντας αντλήσει συμπεράσματα. Είναι σημαντικό λοιπόν να είμαστε μεθοδικοί και ε, να επικρατήσει μια τάξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύω θα καλύψει όλα τα βασικά σημεία αν ακολουθήσει αυτή τη μεθοδολογία για την αξιολόγηση αντικτύπου είναι οι συνήθεις συγκεκριμένοι κανόνες που προβλέπονται, δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω. Ε, ε, συγγνώμη αν παραφθείρω το όνομά σας. Ε, ποιες είναι οι πληροφορίες που πρέπει να ζητούμε για το CBCR, ε, ε, ο τζίρος, ε, ποιο είναι, ποια είναι τα κέρδη, ε, ποια είναι τα ε, φορολογικά βεβαιωμένα ποσά, αυτά που έχουν καταβληθεί. Δηλαδή, θα πρέπει να γίνει αντιστοίχηση ανάμεσα στις οικονομικές δραστηριότητες και τη φορολόγηση χοντρικά. Έτσι θα προχωρήσουμε. Πώς να εφαρμόσουμε την την πρόταση οδηγίας με τον ευρυ... διευρυμένο ορισμό για τις φορολογικές αποφάσεις, τα rulings, Λέμε ότι ζητούνται χωρίς διακρίσεις οι ίδιες ελάχιστες πληροφορίες από όλους και έχουν όλοι ε, την ε, διακριτική ευχαίρεια βάσει αρχής της αναλογικότητας να ζητήσει και άλλες πληροφορίες, ε, επιπρόσθετες πληροφορίες. Επίσης, υποχρέωση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για στατιστική ανάλυση που θα διαβιβάζεται σε όλους. Θα είναι καταλητικός ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε με κάποιο τρόπο να οδηγηθούμε σε μια κύρωση πέρα από τις ε, αποδοκιμασίες κοινή νόμης. Ε, κύριε Ντεμάση, η τωρινή κατάσταση δεν ε, είναι ξεκάθαρη ε, νομίζω ότι αυτή η διαδικασία παραβάση δεν είναι η αποτελεσματικότερη. Εγώ προτιμώ ε, μία πρόταση που θα ενισχύει τις υποχρεώσεις για έλεγχο των κρατών μελών, ε, ε, την, αναβαθμίζει την πρόσβαση στις πληροφορίες και τονίζω επανειλημμένα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα όμως, διότι δεν αποκλείουμε καμία εναλλακτική τη διαδικασία παραβάση. Αν διαπιστωθεί η έλλειψη πληροφοριών, βεβαίω να κινήσουμε τη διαδικασία. Ε, δεν θα διστάσουμε, αυτό προβλέπει και η οδηγία. Ε, εμπιστοσύνη λέτε στις, ε, στους υπουργούς οικονομικών. Γιατί με ρωτάτε, μα στη δημοκρατία η πολιτική ανοίγουν σε μια αιρετή δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση ε, δεν είμαστε και οι καλύτεροι ή χειρότεροι από τους άλλους. Τέλο πάντων υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί, αλλά ε, εκ των προτέρων ε, ε να ε, είστε καχύποπτοι δεν πιστεύω ότι δικαιολογείτε ή άμα θέλετε είναι δικαιωμά σας. Ε, μπορεί κάποιο να μην έχει εμπιστοσύνη του και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί κάποιο να χάσει την εμπιστοσύνη του σε όλα τα θεσμικά όργανα Κύριε Μοσκοβίτση, την κοινή γνώμη μόνο θέλουμε, εμπιστευόμαστε και γι' αυτό ε, ζητάμε νέα διαδικασία. Sorry, can you repeat your... Μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτησή σα δεν άκουσα. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στην κοινή γνώμη που ε, είναι και ειδικοί ε, άνθρωποι και μπορούν να κρίνουν τι σημαίνει ανταλλαγή πληροφοριών. Δηλαδή τι, ε, εννοείται το κοινό, δηλαδή τους ψηφοφόρους ε, και τους ε, ερετούς, ε, δηλαδή το κοινοβούλιο. Ο ε, αγαπητός συνάδελφος Λαμασούρα απάντησε με σαφήνεια. Μέσα από τις εκλογές εκφράζει τη γνώμη του ο λαός. Φυσικά η αντιπροσωπευτική δημοκρατία δεν αντιπροσωπεύει όλους, αλλά Ε, όλοι θα πρέπει να ενημερώνονται και να ε, σέβονται το σύστημα, το οποίο βεβαίως έχει τα όρια του. Γι' αυτό σας ε, είπα ότι η κοινοποίηση έχει μέσα τη λέξη κοινό και για την ενημέρωση του κοινού εγώ θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια. Ως προς την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με το παρελθόν. Καταλαβαίνω αυτή την ερώτηση και μπορώ να σας πω ότι ε, είμαστε νέα επιτροπή. Δεν θα σας το πω όμως. Θα πω πως ε, παλαιότερα βασιζόμασταν στην ε, ανταλλαγή σε θελούσια βάση και δεύτερον, σε αυτόν τον διακυβερνητικό κώδικα δεοντολογίας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όμως διαφορετικά εργαλεία για να εντεπεξέλθουμε στην τωρινή κατάσταση. Δεν έχει όμως αρμοδιότητα στον τομέα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν εγκριθεί η πρότασή της όμως ε, θα ε, προκύψει νομοθεσία και άρα θα μπορούμε να κινούμε διαδικασίες επί παραβάση. Γι' αυτό σας μίλησα για μια μικρή επανάσταση νωρίτερα. Είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά είναι μια ρήξη σε σχέση με το παρελθόν, ε, σε σχέση με την αδιαφάνεια που επικρατούσε το παρελθόν για το Βέλγιο. Βεβαίως υπήρχαν τεκμηρία, αλλά ούτε οι φυστάμενοι κανόνες ε, ήταν ε, σαφείς, ούτε επαρκεί τα πιστήρια και γι' αυτό δεν αναλάβαμε τη δράση που επιθυμούσαμε. Κύριε Ζανή, για την διαφάνεια του Μητρώου δεν το απέρριψα. Είπα ότι στα μέτρα, στο μέτρο του δυνατού αυτό θα κάνουμε και επαναλαμβάνω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ασχοληθεί με την επεξεργασία των πληροφοριών. Α, για την ερώτηση για την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σα ευχαριστώ για την πρότασή σας. Δεν είμαι κατά τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, αλλά σίγουρα θα ξέρετε, διότι είστε υπέρ τη ε, κοινοτική ε, μεθόδου, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει η πλατφόρμα, δημόσια πλατφόρμα για την ε, βέλτιστη διοικητική συνεργασία. Ο κύριο Μονό τώρα ε, είναι φεντεραλιστή ουσιαστικά. Πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι παντοδύναμη και μπορεί να πιέζει τα κράτη-μέλη για να αναλαμβάνει νομοθετικέ πρωτοβουλίε. Σα ευχαριστώ για την υποστήριξή σα, ε, διότι πολιτικό πώ εγώ αυτό το δρόμο ακολουθώ. Ξέρετε όμω ε, υπάρχουν αλλαγέ ε, που γίνονται αθόρυβα και προκύπτουν από συζητήσει που γίνονται και πιστεύω ότι κάποιοι θα με καταλάβουν και θα με υποστηρίξουν για τι αποζημιώσει. Βεβαίω μπορούμε να προετοιμάσουμε εργαλεία ανταλλαγή πληροφοριών. Οι συνέπειε όμω, και πάλι εδώ να πω ότι είναι μάλλον φεντεραλιστική η απάντησή σα, ε, δεν λαμβάνεται υπόψη του ε, ε, ισχύοντε κανόνε που έχουν αποφασίσει τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί παρά να επικροτήσει το φεντεραλισμό σα. Τα κράτη-μέλη δεν, μπορούν, δεν μπορούμε συγγνώμη, να επιβάλλουμε εμεί τα κράτη-μέλη πώ θα κινηθούν σε σχέση με τους, τις επιχειρήσεις τους το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενθαρρύνουμε την ανταλλαγή των πληροφοριών. Είναι ήδη φιλόδοξη η πρότασή μα και επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση ε, και να ακολουθήσουμε πρότυπα παρεμφερή με αυτά που θα θεσπίζει ο ΣΑ. Ε, κύριε Μοσκοβισή, δεν απαντήσατε όμω ε, συγκεκριμένα. Συγγνώμη, διακόπτει ο πρόεδρο Λαμασούρ. πρέπει να ζητήσετε το λόγο αν θέλετε να μιλήσετε. Εντάξει δεύτερος και τελευταίος γύρος ερωτήσεων θα αρχίσουμε με τον πρόεδρο Φέρμπερ που δίνει στον εαυτό του το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ αλλά κύριε Επίτροπε σας ευχαριστώ πολύ για τα όσα μας είπατε. Νομίζω ότι η διαφάνεια είναι σημαντική αφετηρία και κίνητρο, αλλά αφετηρία και κίνητρο γιατί διαφάνεια σημαίνει ότι Ε, ε, το να γνωστοποιούνται κάποιοι κανόνες μέσω της διαφάνειας δεν σημαίνει ότι αλλάζουν κιόλα. Δεν ξέρω αν αρκεί από μόνη της η διαφάνεια. θέτει αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, επειδή είδαμε ότι υπάρχουν μέχρι τώρα 548 τέτοιες συμφωνίες, παρακαλώ. 548 από τα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας. Και αυτό είναι μάλλον μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να διαχειριστούν αυτά οι εφοριακοί στα διάφορα κράτη-μέλη. Πρέπει να το κοιτάξουμε. Δεύτερο. δεν είναι ότι δεν έχει κάνει τίποτα μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 2011 ο προχάτοχό σα είχε κάνει μια πρόταση για κοινή οδηγία ε, για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογία εταιριών. Τον Απρίλιο του 2012 Εμεί νομοδοτήσαμε για το CCTB. Έκτοτε είναι στο Συμβούλιο αυτή η πρόταση. Και ρωτώ, τι προτάσεις θέλετε να καταθέσετε σχετικά, τι, γιατί είναι τόσο κακές οι σημερινές προτάσεις, ε, δεν αξίζει να αναζωογονηθούν. Τι καινούριο θέλετε να φέρετε τον Ιούνιο, αφού υπάρχει αυτή η πρόταση. Και σε μία συνέντευξη στη Βέλτε της Γερμανίας στις 18 Μαρτίου, που σας ρώτησαν για νέους φορολογικούς συντελεστές, αν το φαντάζεστε, είπατε ότι όλα μπορεί κανείς να τα φανταστεί. Αλλά αν δω τις προτάσεις, διαρωτώ με. Ε, αυτό είναι ένα ευρύ φάσμα. Δηλαδή, από την αλλαγή προφοριών μέχρι τους συντελεστέ συντελεστές ε, είναι ευρύ το πεδίο. Ευχαριστώ κύριε Φέρμπερ. Ο κύριο Ραμόν Χαουρέκη, εκ μέρου του SND των Σοσιαλιστών Εκτών. Λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα κύριε Μοσκοβισή καταρχάς να σας πω ότι χαίρομαι και εκτιμώ τη μεγάλη πολιτική σα βούληση στις εργασίες γιατί ακριβώς προβλήματα δεν θα έχετε εδώ στο Κοινοβούλιο αλλά στο Συμβούλιο κατά την απόψή μου. Έχω δύο αμφιβολίες που θέλω να σας διαβιβάσω. Η μία είναι πάρα πολύ βασική. Εντάξει, ανταλλαγή πληροφοριών λέτε και διαβίβαση. Αυτό μπορεί να αφορά οποιαδήποτε εταιρεία, έτσι δεν είναι, ανεξαρτήτως ε, έδρας και εθνικότητας. Είμαι εκπλήσει γιατί διάβασα ε, μία έκθεση του Global Financial Integrity που λέει πάνω από 150 εταιρείες που δεν είναι ευρωπαϊκές και μπορούν να συνδέονται με άλλες χώρες, είναι λέει εκτός της προτάσεως αυτής. Αυτό πώς γίνεται. Είναι λάθος. Έτσι. Θέλω να μου το διευκρινίσετε αυτό, να διαδεσκεδάσετε την αφιβολία. Θα αφορά όλες τις εταιρείες, όχι μόνο τις ευρωπαϊκές. Δεύτερη ερώτηση, η αμφιβολία. Για τις κυρώσεις. Ε, πολύ ωραία τα είπατε. Ε, ωστόσο θυμάμαι εγώ ότι τα κράτη ε, όταν καλούνται να μεταφέρουν τις οδηγίες έχουν κάποιες προθεσμίες και τα λοιπά. Και ανησυχώ για ποιο λόγο. Υπάρχει αυτή η διασυνοριακή ε, διάσταση που είναι και το επιχείρημα που υποχρεώνει τα κράτη-μέλη στην ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτή η διασυνοριακή λοιπόν διάσταση μπορεί να ερμηνευθεί ε, με τρόπο επιλεκτικό. Δηλαδή να μην ενημερώνονται για όλα τα rulings, αλλά μόνο για τα δύο διασυνοριακά, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι ενήμερη για όλες τις φορολογικές πρακτικές όλων των κρατών μελών. Γι' αυτό θα σας παρακαλούσα να θεσπίσετε κυρώσεις σε περίπτωση που τα κράτη-μέλη δεν διαβιβάζουν τις πληροφορίες. Και ένα τρίτο και τελειώνω. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτούς τους καιρούς που οι επιχειρήσεις θέλουν να έχουν καλή φήμη και νοιάζονται για την εικόνα τους και πάνε 10 χρόνια τώρα στην Ευρώπη και παραπάνω. Στην Ευρώπη υποστηρίζουμε την κουλτούρα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων. Οπότε, μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια στιγμή να δημοσιεύει τη σχέση ε, και τις πρακτικές που δεν είναι υπεύθυνες. Αυτό είναι μια υποχρέωση προς το λαό για να έχουν φορολογική υπευθυνότητα και ευθύνη. Ευχαριστώ κύριο Σκύρτσος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, καλωσορίζω και εγώ τον Επίτροπο, ο οποίος έχει αποδείξει ότι ε, στηρίζει την προσπάθεια της Ελλάδας να, να βρει τέλος πάνω την οικονομική, τον, την οικονομική της πορεία. Θα ήθελα λοιπόν να θέσω δύο ερωτήματα ελληνικής αλλά ε, ελληνικής φορολογικής επικαιρότητα με ευρωπαϊκή διάσταση. Το πρώτο ερώτημα. Είναι ε, στην Ελλάδα έχουμε μπερδευτεί με τη φορολογία των εφοπλιστών. Η δική μας κυβέρνηση που, προ... ήταν πριν, η κεντροδεξιά, κεντροαριστερή κυβέρνηση, ήθελε να αποφύγει την αύξηση της φορολογίας των εφοπλιστών, που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο από τη δεκαετία του 50 το δικαίωμά τους να πληρώνουν χαμηλούς φόρους γιατί φοβότανε μήπως φύγουν και πάνε αντί για τον Πειραιά, από τον Πειραιά να φύγουν και να πάνε στη Σαγκάη, στη Σιγκαπούρη. Ε, προσπάθησε λοιπόν να αυξήσει τη φορολογία των Ελλήνων εφοπλιστών σε θελοντική βάση. Τα κατάφερε ως ένα βαθμό και δέχτηκε κοινωνική και πολιτική κριτική, ακόμα και από Γερμανούς συναδέλφους, που λένε ότι πόσο ο Γερμανός φορολογούμενος στηρίζει την ελληνική προσπάθεια με δάνεια τη στιγμή που δεν πληρώνουν οι Έλληνες εφοπλιστές αρκετούς φόρους. Η νέα κυβέρνηση που είναι, έχει, είναι έτσι αριστερή θέλει να φορολογήσει τους εφοπλιστές αλλά και αυτή προβληματίζεται μήπως αυξάνοντας τη φορολογία των Ελλήνων εφοπλιστών που είναι βέβαια πολύ επιτυχημένοι και απόλυτα παγκοσμιοποιημένοι του, τους δει να φεύγουν προς, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης προς ε, Σαγκάη, Σιγκαπούρη ε, υπάρχει, ε, ποια είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορεί, μπορεί να, να αυξήσει τη φορολογία των εφοπλιστών στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να, να, να μείνουν στον ευρωπαϊκό χώρο ή αν προσπαθήσουμε για κοινωνικού λόγους να τους αυξήσουμε τη φορολογία θα τους ψάχνουμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Και το δεύτερο έχει σχέση με την προσπάθεια της νέας ελληνικής κυβέρνησης, που είναι αριστερή, κατά βάση, να έρθει σε συμφωνία με την Ελβετία για να φορολογηθούν οι καταθέσεις εύπορων Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται εκεί, με το Λουξεμβούργο, να δει τι θα γίνει <laughs> με τη γνωστή λίστα Φαλσιανή, που είναι ως γνωστή λίστα Λαγκάρντ στην Ελλάδα. Ε, εν πάση περιπτώσει, το ερώτημα είναι το εξής η, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς αντιμετωπίζει αυτή την προσπάθεια. Θεωρεί ότι θα φέρει συγκεκριμένα έσοδα και τα προεξοφλεί, τα, τα προϋπολογίζει μάλλον για να φτάσει σε μια συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση και να αποδεσμευτούν και οι δόσεις του δανείου και να λειτουργήσει η ελληνική οικονομία ή θεωρεί ότι όλα αυτά θα αποδώσουν σε ένα, δύο, τρία χρόνια οπότε θα τα μετρήσει στο δημοσιονομικό, ναι, στη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος τότε όταν πραγματοποιηθούν και αν πραγματοποιηθούν αυτά τα φορολογικά έσοδα. Ευχαριστώ πολύ. Merci, mon cher Σας ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Ο κ. Κονφεράτη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η άποψή σας σχετικά με το θέμα αυτό της ανάλυσης κατά χώρα όσον αφορά τη φορολόγηση. Έχετε εισάγει κάτι τέτοιο για τις τράπεζες και υπήρχαν φόβοι για αλλίωση του ανταγωνισμού, αλλά ήταν αβάσιμη η φόβη όπως αποδείχθηκε. Λοιπόν, θα ήταν σημαντικό στοιχείο διαφάνειας αυτή η προσέγγιση σε φορολογικό επίπεδο, διότι θα πρέπει επιχειρήσεις στις διάφορες διαστάσεις οποίες κινούνται να δηλώνουν την δραστηριότητά τους κάθε χρόνο και τον φόρο που πληρώνουν στη κάθε χώρα. Σήμερα στο Κοινοβούλιο συζητείται η οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων. Πιστεύω ότι σε αυτή την οδηγία το θέμα της ανάλυσης κατά χώρα της φορολόγησης είναι κάτι που ενδείκνεται και μπορούμε να φύγουμε έτσι από την αμφισημία που κρατούσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έλεγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το σκεφτόμαστε και θα αξιολογήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει συγκεκριμένη δυνατότητα να γίνει κάτι για να ρηχθεί φω όσον αφορά στα μικρά ωφέλη, αλλά ωφέλη που απεκομίστησαν χρησιμοποιώντα ε, αυτό το εργαλείο οι τράπεζε. χρησιμοποιώντα αυτό το εργαλείο για τι τράπεζε. Θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε πιο γρήγορα να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μέσο που είναι στη διάθεσή μας και είναι πάρα πολύ ε, αποτελεσματικό αυτό που είπατε της οδηγίας για τα δικαιώματα των μετόχων. Θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η δική σας άποψη επί της ουσίας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τόμας Μάν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που έχουμε εδώ πολλούς βουλευτές που λέγουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει περισσότερα, να είναι η μεγαλύτερη φιλοδοξία της. Θέλω να θυμίσω ότι εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε κάνει ήδη πολλά. Στην Επιτροπή μας ΕΚΟΝ έχουμε έκθεση πρωτοβουλίας για ε, την κατάργηση των φορολογικών παραδείσων. Μας λένε ότι είναι πολύ ασαφή αυτά και λυρικά. Μα ε, γιατί τα κράτη-μέλη δεν συνεργάζονται. Έχουμε ακούσει υπουργού οικονομικών να συμφωνούν, αλλά συγκεκριμένα βήματα δεν έχουν κάνει. Τώρα θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία, όχι επειδή το απαιτεί η κοινή γνώμη, αλλά γιατί και εμεί, ε, οι βουλευτές το βλέπουμε. Πολλοί μικρομεσαίοι δεν μπορούν να ζήσουν πια, να επιβιώσουν, ε, γιατί πληρώνουν τους φόρους ε, οι μικρομεσαίοι, ενώ οι μεγάλοι αγρίως φοροδιαφεύγουν. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Είναι αφόρητη. Για τη φορολογική βάση, ο Μάρκους Φέρμπερ τα είπε, για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιριών. Είναι δύσκολη. Ε, το ξέρω ότι είναι κυρίαρχα τα κράτη-μέλη, είναι γνωστό αυτό στα φορολογικά, αλλά κάτι πρέπει να γίνει εκεί. Και μετά οι ίδιες εταιρείε. Εγώ αγωνίζομαι εδώ και χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η κοινωνική εταιρική ευθύνη των εταιριών να είναι βεβαίως σε εθελοντική βάση. Αλλά βγάζουν ωραία φυλάδια που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν όμως και συγκεκριμένα γεγονότα και στοιχεία. Ας πούμε, πόση φορολογία, ε, πόσους φόρους πληρώνουν στην κάθε χώρα. Να τα βάζουν και αυτά στα φυλάδια. Και δεν είναι θέμα πολιτικής ευθύνης, αλλά κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. γιατί λέμε ότι δεν υπάρχουν διεθνή πρότυπα. Είναι σωστό αυτό. Ξέρετε ότι είμαι Γερμανός, το ακούτε από τη γλώσσα που μιλάω. Εμείς ε, στο Bundesrat έχουμε μια πρωτοβουλία ε, που θέλει να δημιουργήσει ε, μια δυνατότητα για τις εταιρείες για να λαμβάνουν μια άδεια για τη Γερμανία θα πρέπει να φορολογούνται τουλάχιστον 25% στην άλλη χώρα. Ε, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτά τα παραθυράκια οι μεγάλες εταιρείες ε, για να φοροδιαφεύγουν. Ε, φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει μεγάλη πλειοψηφία στο Bundesrat που εκπροσωπούνται εκεί τα ομόσποδα κράτη να μην υπάρχει πια φορολογικό dumping γιατί τελικά οι μεγάλοι ξεφεύγουν ενώ οι μικροί, οι μικρομεσαίοι, οι εταιρείε μας και οι εργαζόμενοι πλήττονται. Ευχαριστώ κύριε Μπαγιέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που είστε εδώ μαζί μας. Πολλά ήδη υπόθηκαν, αλλά θα ήθελα να επανέλθω συντομία σε κάτι βασικό. Όταν μιλάμε για φοροδιαφύγη, ε, μιλάμε τελικά για την καταπολέμηση αυτή μέσω βελτιστοποίηση φορολογική. Λοιπόν, όταν περνάμε από βελτιστοποίηση φορολογική σε φοροαποφυγή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλε τι τεχνικέ και όλα τα εργαλεία για να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, Ένωση θεωρείται ότι αυτό είναι απάτη οι άλλοι θεωρούν ότι ε, είναι νόμιμο να διαφέρει κανεί από το φόρο, χρειάζεται βελτιστοποίηση τη φορολόγηση. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τι δυνατότητέ μα που έχουμε στη διάθεσή μα. Θα προχωρήσετε επί ενό ορισμού τη φοροαποφυγή και το Συμβούλιο. Δεν μπορεί να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά κάθε χώρα να λέει ορισμό είναι διαφορετικό. Δεύτερον, όταν μιλάτε για φοροδιαφυγή, μιλάμε για επιθετικά συστήματα ε, από συμβούλους, δικηγόρους που χρησιμοποιούν διάφορα, ε, διάφορα συστήματα να ξεφεύγουν εταιρείε από, το από το φόρο. Και έχουν σχεδόν υπερακριβή χαρτογράφηση των διαφόρων νομοθεσιών όσον αφορά τη φορολόγηση των χωρών και έτσι όλοι αυτοί μπορούν να αποφύγουν το φόρο. Αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο, αποτελεσματικά χρησιμοποιήσουμε τέτοια εργαλεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χαρτογράφηση παρόμοια τοπολογικών συστημάτων. Ποιοι κανόνε ισχύουν σε κάθε χώρα. Αν όχι, μήπω δεν ήρθε η ώρα τώρα επίση να γίνει κάτι τέτοιο, να υπάρξει μια μικρή ομάδα ελέγχου και υποπτία, ούτω ώστε κάθε φορά να είμαστε ενήμεροι. Διαφορετικά, αν δεν υπάρχουν τα ίδια εργαλεία από δύο πλευρέ, πώ να καταπολεμηθεί. Τρίτον, σε κάποιε χώρε και στη χώρα μου σύντομα και στον Ηνωμένο Βασίλειο και στι κάτω χώρε κλπ. Για να γίνει, για να πολεμηθεί το φαινόμενο αυτό, το τεχνασμάτι φορολόγηση, έχουν το φόρο καημάν όπω αποκαλούνται για τι επενδύσει που ξεφεύγουν εταιρείε με έδρα στο εξωτερικό. Λοιπόν, ε, ουσιαστικά φορολόγηση αυτή θεωρείται από κάποιε χώρε ότι αντιστοιχεί σε φορολογική αμνηστία. Είναι καλό αυτό ο φόρο Καϊμάν ή ή θεωρείτε ότι είναι φορολογική αμενιστία. Τελευταία ερώτηση τεχνικής φύσεως, αν επιτρέπετε. Που το πρόγραμμα Φισκάλης 2020 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, πώς πάει εδώ και ένα χρόνο έχει ξεκινήσει, οι εθνικές εφορίες έχουν κάνει εναρμόνες των πληροφοριών, είχαν την ευκαιρία να το κάνουν, έχει γίνει αξιολόγηση του προγράμματος, πώς λειτουργεί. Αν όχι, πότε προβλέπετε κάτι τέτοιο. Και τα αποτελέσματα ποια είναι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τόμβαν Κάντελαρ. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, θα μιλήσω Ολλανδικά. Όλοι συμφωνούν εδώ ότι ε, οι LuxLeaks ε, και οι άλλες αθέμητες ε, φορολογικές πρακτικές είναι απαράδεκτες. Για μένα αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να υπάρχουν κοινοί κανόνες για τον υπολογισμό της κοινή ενοποιημένης φάσης φορολογίας εταιριών. Από το 2011, όπως είπαμε, υπάρχει θέση του Κοινοβουλίου, τρία χρόνια είναι στο σιρτάρι του Συμβουλίου και υπάρχει εμπλοκή. Πώς προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απεμπλέξει ακριβώς αυτό το θέμα και ποια είναι τα πιο ακαθόδη ζητήματα. Και θα κάνετε μια τροποποιημένη πρόταση τώρα για να ξεφύγουμε από το εθελοντικό σύστημα σε ένα υποχρεωτικό, όπως ζητούσε και η έκθεση του Κοινοβουλίου. Για τη διαφάνεια υπάρχει μια πρόταση ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ευχαριστώ γι' αυτό. Η διαφάνεια είναι καλή για τα rulings, ε, αλλά όπως λέει και η επιστολή της 28 Νοεμβρίου 2014 που ήταν από τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία, αυτό δεν αρκεί. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο πώς θα γίνουν πιο αυστηροί οι κανόνες ε, για να σταματήσουν τέτοιου είδους συνεννοήσεις και συμφωνίες ε, με τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ. Ε, euh, Καταρχάς προς τον πρόεδρο τον κύριο Φέρμπερ αναφερθήκατε σε στοιχεία, πληροφορίες, τον τύπο κλπ. Άλλοι αναφέρθηκαν στη χαρτογράφηση λοιπόν και ότι πρέπει να υπάρχει κάποια συμμετρία στον αφορά τις πληροφορίες. Ο τύπος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες και μέσω των επιχειρήσεων υπάρχουν ε, πρόσβαση στην πληροφορία. Αυτό που είναι το διακύβευμα είναι ότι την πλευρά του δημοσίου, στο δημόσιο, στο κοινό, να αρθεί η αδιαφάνεια. Θα πρέπει σε επίπεδο επιχειρήσεων και φορολογικών συμβούλων να επικρατεί διαφάνεια. Θα πρέπει μέσω νομοθεσίας να το πετύχουμε αυτό. Αυτό είναι το διακύβευμα των προσπαθειών. Πριν δεν υπήρχαν σαφείς κανόνες. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να προτείνουμε κανόνες σαφέστατους σαν πρώτο βήμα επαναλαμβάνω. Δεν θα περάσουμε από τη σκιά στο φως και από την κόλαση στον παράδεισο. Αυτό που κάνουμε είναι σαφέστατο. Τώρα λοιπόν εξαρτάται από τα κάτι μέλη να θετήσουν τα μέτρα. Το λιγότερο στο οποίο πρέπει να επαγρυπνούμε το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ε, το αναδρομικός χαρακτήρας των μέτρων. Λοιπόν, λοιπόν, αναφερόμαστε σε δεκαετία ε, προύπαρξη των rulings. Συγγνώμη κύριε Επίτροπε. Λοιπόν, πηγαίνουμε πίσω σε δεκαετία για τα ruling που εφαρμόζονται ακόμα σήμερα. Δεν πάμε σε αυτά που έγιναν πριν από δέκα χρόνια και δεν ισχύουν πια. Όπως και το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, κινούμαστε σε αυτά που ακόμα ζουν. Δεν είμαι χριστιανός προσωπικά. Ναι, Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Οπότε δεν διεκδικώ καμία επεράσπιση, καμία θρησκεία, κύριε Πρόεδρε. Δεν με καμία θρησκεία. Λοιπόν, η αναδρομικότητα ε, εφαρμόζεται. Διότι αν εκαλύπτετο, οπότε δεν θα ήταν τόσο αποτελεσματικές οι, κυρώσει. οι κυρώσεις. Όσον αφορά την ενιαία φορολογική βάση κλπ, Ποτέ δεν είπα ότι δεν έκανε τίποτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντιθέτω. Διαδέχομαι το επιτρόπου του κυρίου, τον, τον κύριο Σεμέτα, τον κύριο Επίτροπο που έκανε πολλά πράγματα. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα αυτά που έκανε και τα χαιρετίζω και σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, είναι έξοχη αυτή η, ε, πρόταση, αλλά τι διαπιστώνουμε. Δυστυχώ ότι έχει μπλοκαριστεί το μέτρο στο Συμβούλιο. Δεν θα απαντήσω όσον αφορά το τάξη άμεσα. Ακολουθούμε τη στρατηγική. Θέλουμε να προχωρήσουμε λοιπόν. Εάν η ίδια πρόταση μας επιτρέπει να καταλήξουμε κάποια αποτελέσματα, διότι υπάρχει πολιτική ορίμανση για αποδοχή, θα χαιρόμουν πολύ. Αν ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση, που επιτρέπει να έχουμε ομοφωνία των κρατών μελών, δεν αποκλείεται να κάνουμε κάτι τέτοιο. Τέλος, υποτεθεί στο ότι τίποτα λειτουργεί, υπάρχει δυνατότητα ε, της ε, ενισχυμένης συνεργασίας θα ήθελα όλα τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να εθετήσουν ένα φόρο των εταιριών και των ε, οικονομικών συναλλαγών, ε, διότι αν τα καταφέρουμε στις 28 ε, και δεν μπορούμε ούτε στους 11, δεν θα καταφέρουμε καθόλου. Και γι' αυτό έχουμε ξαναθέσει την πρόταση, να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, το καλοκαίρι λοιπόν, με το πακέτο, το δεύτερο πακέτο, συμφωνήσαμε στατικικά διαβήματα που θα μας βγάλουν από τα διέξοδο και αυτός είναι ο στόχος. Και η βασική πρόταση είναι αυτή που προτιμάστηκε από την προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την υποστηρίζω, είμαι αλληλέγγυος. Να είμαστε ξεκάθαροι στον αφορά αυτό. Ε, ευχαριστώ και Πανή για την υποστήριξή σας. Όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, ναι, όλοι οι φορολογούμενοι, όλοι οι φορολογούμενοι που είναι αντικείμενο ε, ruling καλύπτονται όπως και οι ξένες επιχειρήσεις. Όσον αφορά τις κυρώσεις, από τη στιγμή που ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο παιχνίδι, τα κράτη-μέλη ε, τα οποία δεν συμμορφώνονται θα υποστούν διαδικασία κατά παράβαση. Και προβλέπεται ότι θα επιβληθούν κυρώσεις. Ο κύριος Κίρτσος το γνωρίζει ότι ανεξάρτητα από την ελληνική κυβέρνηση, εδώ και κάποιο χρόνο είμαι ε, ένας που υποστηρίζω την παρουσία της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, την υποστηρίζω, είναι πολύ σημαντικό για τους Έλληνες, για τον ελληνικό λαό και είμαι υπέρ να είναι εμποδιστή η δυνατότητα της Ελλάδας να αναπτυχθεί. Γιατί αυτό είναι το διακύβευμα. Να γίνει πιο ανταγωνιστική, να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και να καλυφθούν και τα προβλήματα, τα δεινά της κοινωνίας ε, των Ελλήνων. Αυτό είναι κοινό διακύβευμα ε, της ε, Ελλάδος, όλων των πολιτικών στην Ελλάδα. Και γι' αυτό εργαζόμαστε εδώ στην Ενώση εδώ και αρκετές ημέρες Γίνονται διαβουλεύσεις μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των εταίρων της. Έχουμε στα πλαίσια της Brussels ε, Group. Εγώ πρότεινα να δημιουργηθεί αυτή. Θα πρέπει να συνεχιστεί και στην Αθήνα επιτόπου η προσπάθεια να βρούμε τα στοιχεία που χρειάζονται με στόχο να λάβουμε υπόψη τις δημοκρατικές προτεραιότητες που χρειάζονται σε μια χώρα από μια δεδομένη στιγμή. Είναι άλλες προτεραιότητες, άλλη στιγμή είναι άλλες προτεραιότητες. Ο λαός επιλέγει αλλά θα πρέπει να σεβαστεί τι υποχρεώσει έναν των εταίρων η Ελλάδα και αυτό είναι θεμελιώδου σημασία. και αυτό σε ένα χρονικό διάστημα μετρημένο, διότι υπάρχουν κάποιε προθεσμίε που πλησιάζουν. Το εργαζόμαστε επ' αυτού, εργαζόμαστε σε καλό πνεύμα και δεν είναι απλά τα πράγματα, δεν είναι εύκολο. Όπω υποσχέζεται δεν μπορώ να δώσω περισσότερε πληροφορίε. Γνωρίζω ότι υπάρχουν ομάδε, παρακολουθώ εκ του σύνεγγυ τη εργασία, που εργάζονται ε, ε, νυχθημερών. Και όταν λέω νυχθημερών, Νυχτημερών εννοώ, κάθε μέρα, κάθε νύχτα και Σάββατα και Κυριακές, όλος ο κόσμος ε, πραγματικά έχει κινητοποιηθεί γι' αυτό. Μετά έχετε θέσει κι άλλο ερώτημα πιο συγκεκριμένο όσον αφορά την φορολόγηση των εφοπλιστών. Δεν, έχουν, δεν μπορώ να απαντήσω αυτό το ερώτημα ίδιος. Είναι, ο λαός τοποθετείται από αυτού, είναι θέμα δημοκρατικό. Θέσατε και τις δύο διαστάσεις του θέματος. Υπάρχει βιολογική διάσταση, ηθική, θέμα δικαιοσύνη. Δεν είμαι Έλληνας. Αγαπώ την χώρα σας. Αλλά δεν είμαι Έλληνας. Και κάποιοι Έλληνες εξέφρασαν με την ψήφο τους κάποια πράγματα. Ε, ε λοιπόν, έγιναν σημαντικές προσπάθειες ε, όσον αφορά εκείνους που είχαν το 27% του ΑΕΠ της χώρας. Γίνανε μεταρρυθμίσεις πάρα πολύ δύσκολε, παραμένουν οι αδικίες, ε, και αυτό είναι απαράδεκτο να υπάρχουν τις ειδικίες και μπορεί να αποτελέσει ε, τμήμα ε, που επηρεάζει ε, την ψηφοφορία στη χώρα. Και μετά υπάρχει το πρόβλημα στην αγωνιστικότητα της χώρας και να μην υπάρχει πρόβλημα φορολογικό. έτσι αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα. Δηλαδή, λαμβάνει υπόψη τις δύο πτυχές. Θέλουμε τη δικαιοσύνη, θέλουμε τη διαφάνεια. θέλουμε ηθικο, την ηθική. Είναι θέματα διντολογικά που τίθενται. Και από την άλλη πλευρά δεν θέλουμε η επιχειρηματική διαστηριότητα να αποδυναμωθεί. Τι νόημα έχει η δεντολογία και η ηθική και η δικαιοσύνη αν δεν δημιουργείται πλούτος. Γιατί λοιπόν να μην ισχύσουμε λοιπόν τους κανόνες με τη διαφάνεια, με πιο στοχευμένους φόρους, αλλά η ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών πρέπει να εδράζεται πρακτικών διαφανών, μη επιζημίων και σε αυτό το πλαίσιο ε, αυτή η προσπάθεια καταβάλλεται που δεν είναι απεχθής αλλά πρέπει να εφαρμόζεται με διακριτικό τρόπο. Γι' αυτό συνετά κινούμε και δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά όταν απαντάω στην ερώτησή σας. Το ίδιο ό, όσον αφορά ε, με την Ελβετία συνεχίζεται ο διάλογος μεταξύ των ελβετικών και ελληνικών αρχών. Θα προτιμούσαμε σφαιρική και συντονισμένη προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά εξαρτάται τα κράτη-μέλη να εξετάσουν και τις διμερείς πρωτοβουλίες τους και στο φορολογικό τομέα και με αυτόν τον τρόπο να προσεγγιστεί το θέμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά το, θέμα, το ερώτημα του κυρίου Κονφεράτη, θα δράσουμε, σα το εγγυώμαι αυτό, ε, δεν είμαι εδώ να λέω ότι δημιουργούμε μια επιτροπή για να θάψουμε ένα πρόβλημα. Κάποιο πολιτικός άντρα από την περιοχή μου ή κάποιο άλλο από άλλη περιοχή το έλεγε αυτό. Ο Ρίκο Έγιο Γκαρφόρ το έλεγε. Κάποιοι πολιτικοί άντρε της δημοκρατίας με ιδιαίτερε παραδόσει χρησιμοποιούσαν αυτή την προσέγγιση. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να γνωρίσουμε πώ θα δράσουμε. Λοιπόν, γι' αυτό δεσμεύομαι εδώ. Να αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα το πρόβλημα, εθελοντικά, για να βρούμε μια λύση. Δεν θέλω να χρονοτριβούμε. Και γι' αυτό με μεγάλη προσοχή παρακολουθώ τι τοποθετήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την οδηγία για του μετόχου, συνεργασία με τον συνάδελφο Ιλ. Λοιπόν, όταν μιλώ για μελέτες αντιχτύπου δεν είναι για να θάψουμε το θέμα αλλά για να δράσουμε συγκεκριμένο τρόπο, στοχευμένο τρόπο με στόχο την ανταγωνιστικότητα. Όχι για απλή ικανοποίηση και ε, για να είμαστε επιβλαβείς για τις επιχειρήσεις. Είμαι υπεύθυνο για την φορολογία. Μπορούσα να αναφέρω και άλλους συναδέλφους. Λοιπόν, υπάρχει γενικώ μια ευαισθησία για το θέμα. Θέλουμε να συνδυάσουμε τα διάφορα στοιχεία που απαιτούνται. Όσον αφορά τον κύριο Μαν, ε, είμαι πολύ κοντά στις θέσεις που έχετε. Όσον αφορά τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, καταλαβαίνω την άποψή σα. Είναι ένα θέμα ισότιμη αντιμετώπιση, ε, των σεβασμού των κοινωνικών συμβάσεων. Ε, λοιπόν, και η θέση μου είναι πολύ κοντά σε αυτά που είπατε εσεί στη δική σα θέση. Όσον αφορά τα τεκτενόμενα στην Γερμανία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει για μια εφαρμογή ε, των κανόνων περί μη καταχρήσεων στο εθνικό επίπεδο και ε, συμφωνώ με τι προσεγγίσεις χώρας. Ο κύριος Μπαγιέ μου έθεσε μια ερώτηση για βελτιστοποίηση και αποφυγή των φόρων. Είναι θέμα νομικό. Νομικής βάσης ή μη νομικής βάσης των συστημάτων. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα δύο φαινόμενα με διαφορετικά εργαλεία ίσως. Δεν μπορούμε να αφήσουμε να μην υπάρχουν κέρδη που δεν φορολογούνται καθόλου στα πλαίσια των διαδικασιών που προτείνουμε, των προτάσεων που κάνουμε, που αφορούν τη διαφάνεια, πρόκειται περί ruling και μετά έρχεται η διαφάνεια και θα ασχοληθούμε και με τη βελτιστοποίηση, τη φοροδιαφυγή, την φοροαποφυγή. Θέλαμε μια μέθοδο διαφανή παρά μια και ένα περίπλοκο νομικό ορισμό ε, που θα ήταν πολύ δύσκολο να εφετηθεί από τα κράτη-μέλη. Βέβαια, κάποιοι θα μας πείτε και το λέτε, το ξέρω ότι εσείς δεν απαγορεύετε, δεν ορίζετε. Όχι. Θέτουμε ένα μηχανισμό, θεσπίσουμε ένα μηχανισμό διαφάνειας που πιστεύω ότι είναι ηθικός, ότι είναι δίκαιος και για μία ακόμη φορά προβλέπονται διαδικασίες ε, που μπορούν να οδηγήσουν οι διαδικασίες σε κάποιες παραβάσεις και θέλουμε να έχουμε αποτρεπτικά μέτρα στον φάτη προσέγγιση, στον φάτη χαρτογράφηση που αναφέρατε, ε, γνωρίζουμε τις δυνατότητες ε, που δημιουργούνται από τις διαφορές όσον αφορά τα φορολογικά συστήματα δεν έχουμε κατάλογο, δεν έχουμε χάρτη, δεν έχουμε διαγράμματα και σήμερα οι επιχειρήσεις και οι φορολογικοί σύμβουλοι είναι πιο δυνατοί από εμά, εξορισμού, διότι εκείνοι ε, ε, έχουν πιο άμεση επαφή και φορολογούνται άμεσα, ενημερώνονται για το ποσοστό τη φορολόγηση και ενημερώνονται και εκμεταλλεύονται ενδεχόμενε τρευλώσει. Λοιπόν, απαντώ στι ερωτήσει Εγώ δεν έχω αμέσω μία απάντηση να σα δώσω αυτά που είπατε. Όσον αφορά το ερώτημα του κ. Βαντεντίντελερ, όσον αφορά το αξί και τον ε, την φορολογική βάση, αν υποχρεωτικό χαρακτήρα ή όχι. Λοιπόν, είναι μία από τι παραμέτρου που εξετάζουμε Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι το σύστημα θα είναι εφαρμόσιμο από τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν να εμπιστευτούμε τα κράτη-μέλη όσον αφορά τις συναλλαγές τους. Θα ήταν δυνατό να υπάρχει διαφάνεια μέσω των φορολογούμενων σας συλλέγουμε από τις πληροφορίες. Και κλείνω από αυτού. Αυτό που προτείνουμε πιστεύω ότι είναι επαναστατικό διάβημα, είναι καινούριο, ανοίγει ένα μονοπάτι, αλλά δεν καταλήγει κάπου, δεν είναι τελικός στόχος και δεσμεύομαι να προχωρήσουμε περισσότερο. Η διαφάνεια ε, είναι το κοινό ε, που αφορά όλα τα επαγγέλματα, όλες τις χώρες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να μπορούμε να συνεργαστούμε από αυτού ε, και περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον όλες τις εργασίες, όλες τις προτάσεις θα κάνετε. Σας το είπα κύριοι Πρόεδροι ότι είμαι έτοιμος να επανέλθω οποιαδήποτε στιγμή τώρα που άνοιξαν οι συζητήσεις και ανα οποιαδήποτε στιγμή μπορούν γραπτώς να απαντήσουν οι υπηρεσίες ερώτημα που μπορεί να υποβληθεί από την Επιτροπή σας, τις Επιτροπές σας για τα θέματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κοντά στο Κοινοβούλιο όσον αφορά αυτά τα θέματα, σας το κρύβω. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ε, τα μέλη μας είχαν την ευκαιρία να θέσουν όλες τις ερωτήσεις που επιθυμούσαν να υποβάλουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ που απαντήσατε με τόσο συγκεκριμένο τρόπο. Συχνά βλέπουμε τη σύγκριση το μισό γεμάτο ή μισό άδειο ε, ποτήρι. Εδώ έχω ένα άδειο μπουκάλι και ένα μισό γεμάτο. Κοιτάξτε, για μας ποιο είναι το θετικό στη δική μας δράση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε το ίδιο, τον ίδιο στόχο τελικά. Και είμαστε σε ένα αγώνα δρόμου. Ε, έχουμε μια άμυλα, ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τον ίδιο στόχο και το μέγα πολιτικό εμπόδιο που έχουμε μπροστά μας, το αναφέρατε πολλοί από εσά, είναι οι κυβερνήσεις και συγκεκριμένα τα Υπουργεία Οικονομικών. Οι μεν διότι επιθυμούν να διατηρήσουν την κάπως προνομιούχο θέση που έχουν και οι δε επειδή είναι κλιμαζοχιστές δεν θέλουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ανακατεύονται με τα εθνικά του ζητήματα. Εμείς θα παραμείνουμε αυστηρά στις αρμοδιότητες και τις εξουσίες της Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στα φορολογικά ζητήματα είναι πάρα πολύ περιορισμένα, ειδικά δε του Κοινοβουλίου οι αρμοδιότητες. Έχουμε όμως πολιτικές ευθύνες. Σημειώνω ότι στο έγγραφο για τη διαφάνεια που είναι το πρώτο στοιχείο της δέσμης που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από λίγες μέρες, ένα από τα βασικά σημεία θα είναι το εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι αποδέκτης των πληροφοριών που θα διαβιβάζουν τα κράτη-μέλη το ένα στο άλλο υποχρεωτικά. Γιατί εκεί είναι το κλειδί των ενδεχομένων κυρώσεων. Κατανοούμε ότι δεν θα ξετρελαθούν όλα τα Υπουργεία Οικονομικών από τον ενθουσιασμό τους όταν το μάθουν αυτό. Επίσης σημειώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει θετικά την ιδέα να δημοσιεύονται υποχρεωτικά οι πληροφορίες ανά χώρα. Βέβαια εκτιμώντας πάντα τις πρακτικές συνέπειες που αυτό θα έχει. Αλλά η Επιτροπή ΕΚΟΝ είχε συμφωνήσει και τέθησε ισχύ για τις τράπεζες. Ήδη εφαρμόζεται αυτή η υποχρέωση, για ποιο λόγο να μην επεκταθεί και αλλού. Επίσης, θα πρέπει θετικά να δούμε τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να προτείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι υποδειγματική στην εφαρμογή των συστάσεων του G20 και του όσα. και πιστεύω ότι δεν διαστρεβλώνω τα λεγόμενά σας, ούτε προδίδω τίποτα. Μας αναγγείλατε ότι τον Ιούνιο θα φέρετε τις προτάσεις ουσιαστικές και αν κατάλαβα καλά θα έχει και νομοθετικές ρυθμίσεις και σχέδιο δράσης σε άλλους τομείς. Συνοψίζω λέγοντας ότι είναι όλες οι προτάσεις του ΩΣΑ αλλά όχι μόνο του ΩΣΑ, γιατί εμείς είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε εσωτερική ενιαία αγορά με πολλά κράτη-μέλη και σε λίγα χρόνια όλα τα κράτη-μέλη θα έχουν νέο νόμισμα. Άρα είναι φυσιολογικό να έχουμε δικούς μας κανόνες, ειδικού. Θετικά λοιπόν όλα αυτά και όπως είπατε αυτή είναι η πρώτη μόνο ακρόαση θα ακολουθήσουν και άλλες. Ε, θα έρθει η κυρία Βέσταγκερ, η Λετωνική Προεδρία επίσης. Και τώρα στη συνέχεια συνεδριάζουν οι συντονιστέ για να εκπονήσουν το πρόγραμμα εργασιών μας. Και έρχομαι να προσθέσω το εξίσου. Σήμερα μας ετοίμησε με την παρουσία της η πρόεδρος της Ολλανδικής Βουλής οι συντονιστές υποστηρίζουν και εκείνη την πρόθεση που έχω να προτείνουμε σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια όσο το επιθυμούν να συνεργαστούμε στενά για αυτό το θέμα. Ο κύριος Ντεμάζη μίλησε για την κοινή γνώμη. Ε, αυτό που χρειαζόμαστε για να αυξηθεί ο πολιτικός αντίκτυπος των προτάσεών μας και κατά κάποιο τρόπο η νομιμοποίηση ε, τους έχουμε ανάγκη να ε, στηριζόμαστε και στα εθνικά κοινοβούλια και τα όσα πράττουμε εδώ να τα λαμβάνουν υπόψη και να τα ακολουθούν και να συμφωνούν μαζί μας μετά από συνεννόηση οι εθνικοί βουλευτές. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, εδώ εξαντλείται η μερίσια διάταξή μας. Ραντεβού αύριο σε άλλη κοινή συνεδρίαση υπό την ηγεσία της ΕΚΟΝ και σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Τάξη, επόμενη συνεδρίαση έχει προβλεφθεί για τις 16 Απριλίου. Διακόπτεται η συνεδρίαση. Παρακαλώ όσοι δεν συμμετέχουν στη συνεδρίαση των συντονιστών να αποχωρήσουν. Μέσα σε λίγα λεπτά και αμέσω μετά ακολουθούν συντονιστές. Ευχαριστώ.